Ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. We can slowly... Να αρχίσουμε σιγά σιγά. Με χαρά, εξ ονόματος όλης της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, Καλωσορίζω τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και σήμερα θέμα συζήτησης είναι ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση από τον κύριο ε, Γιώργη Τόμετ για τα αποτελέσματα της ε, υπουργικής διάσκεψης ε, της δικού σας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ε, με ημερομηνία διεξαγωγής την 17η ε, Νοεμβρίου, όπως έγινε και το, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με σύνθεση και πάλι Υπουργών Εξωτερικών. Ε, νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας από τότε που αναλάβατε καθήκοντα και νομίζω ότι ε, έχουμε πολύ περισσότερα να συζητήσουμε και θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε και στα επόμενα χρόνια. Κύριε Ντόμεκ, έχετε το λόγο για να μας ενημερώσετε για την σε αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά μου πάντα να έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας για να σας ενημερώσω για τις δραστηριότητες του οργανισμού μας. Ε, μακάρι να μπορούσα να σας μιλήσω από καλύτερες συνθήκες. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να τονίσω ότι αντιμετωπίζουμε μια εντελώς νέα πραγματικότητα σήμερα. Ε, ως αποτέλεσμα των τραγικών γεγονότων στο Παρίσι, στη Γαλλία, έχει ε, γίνει πλέον εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απάντηση σε επιθέσεις. Αυτό ήταν ε, πρωτοφανές. Την περασμένη εβδομάδα οι Βρυξέλλες ήταν σε πλήρη αποκλεισμό και υπό τον υψηλότερο συναγερμό που σημαίνει ότι ε, πρόκειται για άμεσο κίνδυνο. Ε, το θέμα είναι ότι πραγματικά χρειαζόμαστε γεγονότα σαν το Παρίσι για να μας αφυπνίσουν. Πραγματικά χρειαζόμαστε ε, άμεσες απειλές ε, στο εσωτερικό μας πριν ε, δράσουμε και προχωρήσουμε με την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ελπίζω πραγματικά ότι όχι. Χρειαζόμαστε τις κατάλληλες δυνατότητες, μια υγιή ε, πολιτική εξοπλισμών που θα υποστηρίζει και τις αμυντικές βιομηχανίες μας, ενισχυμένες συνέργειες πολιτικού στρατιωτικού σκέλους και σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για να κάνουμε αυτό το κβαντικό άλμα. Ε, το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού μας στις 17 Νοεμβρίου ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά. Πριν ε, σας ενημερώσω λοιπόν για τα αποτελέσματα του Διοικητικού Συμβουλίου και ε, σας πω δύο λόγια και για το μέλλον του οργανισμού μας, θα ήθελα να αφερθώ στην παγκόσμια στρατηγική πάντα ε, επισημαίνω δύο ουσιαστικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει κάπως να αντανακλούνται στη συνολική στρατηγική μας. Καταρχάς, ε, στην ανάγκη να αναπτύξουμε τις κατάλληλες δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεύτερον, την ανάγκη να υπάρχει μια ισχυρή ε, ευρωπαϊκή βάση αμυντικής ε, άμυνας και βιομηχανίας και τεχνολογίας και να διασφαλίσουμε και την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αφορά τις βιώσιμες δυνατότητες να αναπτύξουμε, να τροποποιήσουμε και να επιχειρήσουμε ε, σε διαφορετικά πλαίσια. Όταν ε, απίθυνα το λόγο στην ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έμεινα πριν από τρει εβδομάδε. Η ύπατη εκπρόσωπο ε, επεσήμανε την ανάγκη να αναπτύξουμε ένα έγγραφο με σαφέ ε, στρατιωτικέ απαιτήσει. Αυτό θα μπορούσε να πάρει την ε, μορφή μια υποστρατηγική και η μελλοντική Ολλανδική Προεδρία θα καταρτήσει ένα έγγραφο για τις προτεραιότητές μας θα ορίτε δεδομένο βεβαίω ότι ο Οργανισμός Άμυνα θα πρέπει να συμμετέχει και στην, ε, ε, σε άλλους, ε, μαζί με άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα την υπηρεσία εξωτερική δράση. Θα πρέπει επίσης το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωση για την άμυνα να ενισχύσει την ενιαία αγορά για την άμυνα και να απαντάσει σε τέτοιε ε, ανάγκες δυνατοτήτων. Επομένω, θα πρέπει να υπάρχει σαφή σχέση με το πρόγραμμα δράσης και θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ορισμός ε, του ε, βιομηχανικού τομέα άμυνας με βάση τις δυνατότητε που χρειαζόμαστε. Περαιτέρω, Χρειαζόμαστε και κάποια υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία θα ανακύψουν όταν θα αρχίσει να διαμορφώνεται η παγκόσμια στρατηγική. Θα πρέπει να καθαρίσουμε σαφώ ποια είναι τα ε, μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Για παράδειγμα, σε ποιο βαθμό θα επικεντρωθούμε σε δυνατότητε που σχετίζονται με επιχειρήσει ε, ε κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και σε ποιο βαθμό και σε ποιο ε, εύρο θα ληφθούν υπόψη. Σε αυτό το σημείο η πολιτική συζήτηση για το τι ακριβώς περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι ακόμα εν εξελίξη και φυσικά η Ολλανδική Προεδρία θα μπορούσε να συνεισφέρει στη συζήτηση αυτή με τα κράτη-μέλη. Βεβαίω έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι ποτέ να γίνει με τεράστια προσπάθεια και με τεράστιο άλμα ε, στη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Ε, προσβλέπω λοιπόν στο αποτέλεσμα της Συνόδου της Βαρσοβίας, ε, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεάσει τις ενεξελίξει εργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ανάπτυξη των βασικών στόχων, για παράδειγμα, των headline goals, ε, από την άλλη, από πλευρά ΝΑΤΟ, η σύνοδο του ΝΑΤΟ κατά πάσα πιθανότητα θα μα δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια ω προ ε, ε, το Framework Nations Concept. Το αποτέλεσμα λοιπόν τη Βαρσοβία θα πρέπει να συμπεριληφθεί σαφέστατα στο έργο μα ε, στον οργανισμό. Τώρα, ε, προβλέπω ήδη ότι το θέμα του hybrid θα ανακύψει περισσότερο από ό,τι ποτέ ως κεντρικό σημείο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και προς τις δύο κατευθύνσεις. Τέλος, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό το σημείο, πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε να έχουμε το λεγόμενο καταμερισμό αρμοδιοτήτων, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πιεστεί στην γωνία των πολιτικών αποστολών της ήπιας δύναμης και το ΝΑΤΟ θα αναλάβει τις ε, ε, αποστολές υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι πλέον έχει γίνει απόλυτα σαφές ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν συνάδει καθόλου με την έκκληση της Ευρώπης να επενδύσουμε περισσότερα στην άμενα, να παρέχει η ίδια την ασφάλειά της και να είναι πάροχος ασφάλειας και όχι καταναλωτής ασφάλειας και να παραμείνει τελικά ένας σημαντικός παγκόσμιος παράγων. Εδώ έρχομαι και στο δεύτερο ε, στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, τα αποτελέσματα της ε, Υπουργικής Διάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου. Θα ξεκινήσω με τα βασικά προγράμματα δυνατοτήτων του οργανισμού μας. Ο οργανισμός ε, δεσμεύεται ενεργά για την υποστήριξη των τεσσάρων βασικών παραγραμμάτων... που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2013 ε, ανεφοδιασμό air to air, ε, τα ARPAS, ε, τα τηλεκατοφαινόμενα αεροσκάφη, τα drones, το GovSatcom και, το και την κυβερνοασφάλεια, την κυβερνοάμυνα. Τώρα, οι δυνατότητε για το European Strategic Tag. Ε, στόχος μας είναι, υπό την ηγεσία των Ολλανδών, να υπάρξει υπογραφή της σύμβασης ε, το 2016 και το ενδιάμεση αναθεώρηση στα μέσα του 2020. Στόχος είναι να διευκολύνουμε τη συμμετοχή επιπλέον κρατών μελών, να επιτύχουμε συνέργειες ε, στην υποστήριξη με αντίστοιχου στόλους στην Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία και στην κατάρτιση. Και ε, να συνεχίσουμε επίσης για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που διαθέτει ήδη η Ευρώπη ή θα διαθέτουν στο εγγυ μελλον μέλλον. Τώρα, air-to-air refueling ε, θα γίνουν αξιολογήσει εδώ συμβατότητας ε, στα Ιταλικά και η C767 και επίσης θα γίνουν και σε άλλα τάνκερ όπως το Α33 MRTT και το KC46 για να υπάρχουν άδειε σε όλους τους Ευρωπαϊκού δέκτε για το AAR. Επίσης, ε, γίνεται κατάρτιση για τάνκερ και ασκήσεις και υπάρχει ένας διάλογος με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη χρήση των ε, ε, εναλλακτικών δυνατοτήτων Voyager. Επίσης, σκοπεύουμε να βελτιστοποιήσουμε το Α400M ως πλατφόρμα τάνκερ και θα αξιολογήσουμε και τη συμβατότητα Air-to-Air. European Airpass, ένα πρόγραμμα τεσσάρων κρατών, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, υπό την ηγεσία της Γερμανίας στόχος είναι να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα Mailer Pass, το οποίο θα ξεκινά με μια μελέτη καθορισμού, το οποίο θα ξεκινήσει στα τέλη του 2015 και από εκεί και πέρα να διευκολύνουμε τη διάδραση με άλλους πιθανούς εταίρους κατά την ε, φάση της ανάπτυξης. Ο οργανισμός μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνουν τις προσπάθειές τους ε, στον τομέα της, ε, των αεροπορικών μεταφορών, την πιστοποίηση και τον κανονισμό για την ασφαλή ένταξη του ΕΡΠΑΣ στο ε, κοινό εναέριο χώρο. Ο στόχος είναι να εναρμονίσουμε το ΕΡΠΑΣ και τις απαιτήσεις ε, αεροπλοείας μεταξύ των κρατών μελών. Και τέλος, η EDA εργάζεται προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη απαιτήσεων, λειτουργικών απαιτήσεων διπλής χρήσης για το ΕΡΠΑΣ στο ευρύτερο πλαίσιο του ενιαίου ουρανού. Ε, θα υπάρχουν πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του πλαισίου που παρέχει επιχειρησιακή ασφάλεια για το ΕΡΠΑΣ. Επίσης θα υπάρξουν ε, και θέματα που βασίζονται σε προδιαγραφές διετής χρήσης και κανονισμούς και θα αναπτύξουμε δυνατότητες αγορές ε, για τις πολιτικές πτυχές του Ευρωπαϊκού ΕΡΠΑΣ και θα δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος για την ανάπτυξη και την παραγωγή. Ο οργανισμός μας ε, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου, το ΣΕΖΑΡ και τη Eurocontrol, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε δυνατότητες για διπλή χρήση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που θα υποβληθούν στα κράτη-μέλη για περαιτέρω ένταξη στο ΣΕΖΑΡ. Το GovSatcom, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2013, ανέθεσε στα κράτη-μέλη με την υποστήριξη του οργανισμού μας και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ε, Οργανισμό Εξωτερικής Δράσης και τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας να προετοιμάσει την επόμενη γενιά του GovSatcom για το πλαίσιο του 2015. Ε, θα υπάρχει και στρατιωτική και πολιτική σκοπιά και θα καλύψουμε δύο ε, σύνολα αναγκών που θα συγκεντρώσει ο οργανισμός μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, έχουμε το πιο προσαρμοσμένο σύστημα. Έτσι θέλουμε να έχουμε βασικές προτάσεις προγραμματικές οι οποίες θα λάβουν σαφές υπόψη τους τη διπλή χρήση καθώ επίση την ασφάλεια εφοδιασμού, την καινοτομία και την υποστήριξη προ την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και γι' αυτό ακριβώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σωστά θέματα διαχείριση και να αποφύγουμε την κατάσταση που είχαμε σε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, τα οποία δεν είχαν προβλεφτεί αρχικώ ω διπλά ε, και δημιουργήθηκαν δυσκολίε με τις ε, δυνατότητε άμυνα και ε, δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, όπω για παράδειγμα τον Καλλιλέο και τον Κοπέρνικο. Ε, το θέμα της εποπτείας του διαστήματος και της, ε, του εντοπισμού απέδειξε ότι υπάρχει δυνατότητα να συμφιλιώσουμε τις δύο πτυχές και αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα θα πετύχει μόνο όταν τα κράτη-μέλη, ο Οργανισμός Άμυνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας θα μπορέσουν να επινοήσουν τρόπους για να συνεργαστούν με, σε ένα ευαίσθητο και περίπλοκο θεσμικά πλαίσιο. Τώρα, κυβερνοασφάλεια. Δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευση, της κατάρτιση ε, και των ασκήσεων, ε, τον ανθρώπινο παράδειγμα, τεχνολογίες και συμπληρωματικέ με την πρωτοβουλία EUMS για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Υπάρχουν προγράμματα ad hoc ε, για τα διάφορα κυβερνοπρογράμματα ε, και υπάρχουν, ε, θα εγκρίνουν, εγκρίθηκαν μάλλον τον Ιούνιο του 2015 οι βασικές απαιτήσει ε, προσωπικού και τα βασικά στοιχεία για το πρόγραμμα και είναι εν και θα υπογραφούν το Μάρτιο του 2016. Και επίσης υπάρχει το ε, διάφορα πακέτα Cyber Defense Situational Awareness ε, για τις έδρες ε, για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί προς έγκληση τα, οι απαιτήσει για το προσωπικό. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε τα πρώτα project υπό την αμπρέλα του JIP το 2017. Το JIP θα μας επιτρέψει να ενοποιήσουμε υπό ένα οργανισμό όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την άμυνα στον κυβερνοχώρο καθώς και την τα κυβερνητικά και τα βιομηχανικά μέρη, σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά συνεργατικά προγράμματα, το Διευθύνων Συμβούλιο έχει υποστηρίξει το ρόλο του οργανισμού να προωθήσει τις προσπάθειες συνεργασία, ε, ακολουθώντας μία προσέγγιση από πάνω κατά κάτω και βάση ε, του προγράμματος, του αναπτυξιακού προγράμματος ικανοτήτων. Η έρευνα έχει ερευνήσει και προτείνει στα κράτη-μέλη πιθανές δραστηριότητες ικανοτήτων για το μέλλον. Γι' αυτό το σκοπό αρχικοί οδικοί χάρτες έχουν εκπονηθεί για το BioJ Deal, ε, για την Υγειονομική Εκένωση και για ε, τα αντιαρματικά που καλωσορίστηκαν από το Συμβούλιο στις 17 Νοεμβρίου η ε, έγκαιρη αποκλιμάκωση με το ΝΑΤΟ ήταν και θα συνεχίσει να ε, είναι αντικείμενο επαφών σε σχέση με άλλα πιθανά project για την ε, εναέρη υποστήριξη διαθελάσεις και για την ναυτική επιμελητία. Θα συνεχίσουμε να ευθυγραμμίζουμε τη δραστηριότητα και να λαμβάνουμε απόψη τις στρατηγικές επισκοπήσεις ε, προκειμένου ε, να συζητηθούν στο Συμβούλιο όταν θα είναι όριμες. Τώρα να σας πω ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από τους χάρτες. Γιατί επιλέξαμε αυτούς τους τομείς. Καταρχήν ε, υπάρχουν ελλείψεις προτεραιότητες που προέρχονται από τον επιτεξιακό σχέδιο ικανοτήτων δεύτερων απαιτήτων από ουσιαστική μάζα ενδιαφερομένων κρατών μελών, 8 έως 12 αναπερίπτωση τρίτων μπορούν να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και τέλος και συνεχίζω να επιμένω σε αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δεν είναι μόνο σε οργανισμός μεγάλων προγραμμάτων. Όταν μιλάμε για συνεργατικά προγράμματα άμυνα. Θα πρέπει να παραπέψουμε στο έργο που κάνουμε για τη συνεργασία. Επίση, η έρευνα και ε, η τεχνολογία και η απόκτηση εξοπλισμού πέφτουν από το 2006. Έχουμε μείωση 8%. Έτσι λοιπόν πρέπει να δράσουμε όπου είναι δυνατό μέσω τη υιοθέτηση τη αναθερωμένης απόφασης ε, η εξαίρεση από το ΦΠΑ είναι πραγματικότητα. Η εξαίρεση από το ΦΠΑ θα εφαρμοστεί όπου υπάρχει σαφή προσθεμένη αξία του οργανισμού και θα συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να εντοπίσουμε ευκαιρίες να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης προχωρούμε το έργο μα σε χρηματοοικονομικά κίνητρα και θα αναφέρω ε, σχετικά όταν έχουμε αποτελέσματα. Επίσης, ξεκινάμε ένα μηχανισμό ανταλλαγής. Ε, ουσιαστικά πρόκειται για μια πιο εκτεταμένη πρακτική από ότι θα ανέμενε κάποιο ένας τέτοιος ε, αποτελεσματικό μηχανισμός ανταλλαγή στην Ευρώπη θα διευκόλυνε την ε, ανταλλαγή ή τον επιμερισμό ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών με ένα τρόπο αποτελεσματικό του κόστους. Ε, θα κάνουμε ε, ένα εγχείρημα αποτίμησης στο πρώτο εξάμεινο του 2006 και θα θέσουμε προτάσεις στα κράτη-μέλη κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2016. Τώρα έρχομαι στο hybrid. Ο Οργανισμός Άμυνας θα προβεί σε υβριδικές ασκήσεις το Φεβρουάριο και τον Ιούλιο του 2016 με στόχο να προβεί σε δοκιμές των στρατιωτικών ικανοτήτων σε ένα περιβάλλον υβριδικής απειλής. Έτσι λοιπόν αυτό θα διευκολύνει την αξιολόγηση των συνεπειών του υβριδικού πολέμου για τις υφιστάμενες ικανότητες και θα συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Κομισιόν και το ΝΑΤΟ. Ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμένα σε ένα κοινό πλαίσιο ε, για την ε, αντιμετώπιση των ε, υβριδικών απειλών και συνεισφέρουμε σε μια δραστηριότητα που διεξήθηκε στο πλαίσιο της εξαιρετίας 2015-2016. Και φυσικά βελτιώνουμε και τη συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ που σας ανέφερα. Σε ό,τι αφορά την έρευνα και την τεχνολογία, η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης πρέπει να υποστηρίζεται από πολιτικές εργαλεία και επενδύσεις σε στρατηγικές δραστηριότητες κλειδιά. Χρειάζεται λοιπόν προτεραιότητα να θέσουμε σε προτεραιότητα τις προσπάθειες και μία προσέγγιση εφιούς επένδυσης από τα κράτη-μέλη. Ε, η προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα που σχετίζεται με την ΠΑ μπορεί ουσιαστικά να αλλάξει το παιχνίδι για να νομολογήσει μελλοντική έρευνα και ένα πρόγραμμα άμυνας. Το μέρο του 2015 ε, το Συμβούλιο επικύρωσε τις ε, απόψεις των ε, Υπουργών Άμυνας για την διαχείριση και τους τρόπους της προπαρασκευαστικής δράσης. Η ομάδα των προσωπικότητων που δημιουργήθηκε από την Κομισιόν θα εκπονήσει μία Έκθεση για του στόχου, τι συστάσει, τη διαχείριση και του τρόπου του Φεβρουαρίου του 2016. Ο οργανισμό συνεχίζει να συνεργάζεται με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη με μία σειρά workshop για να διευκρινίσει πώ μπορούμε να λάβουμε καλύτερα υπόψη τι ιδιαιτερότητε τη έρευνα στην άμυνα. Η Κομισιόν, η DA και οι νομικοί προγνώμονε των κρατών μελών του επόμενου ε, μήνε ε, θα συναντηθούν σε ομάδες εργασίας. Επίσης, θα επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο και στη χρήση των εφιστάμενων μηχανισμών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για να εντοπίσουμε τις ικανότητες και τις προτεραιότητες έρευνας. Όπως γνωρίζετε, με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση του 2015 επίση προέβλεπε ένα πιλωτικό πρόγραμμα με δύο δραστηριότητε στον τομέα τη ε, αμυντική έρευνα. Ε, η απαραίτητη συμφωνία μεταξύ τη Κομισιόν και τη CDA υπεγράφει στι 16 Νοεμβρίου. Η μεταφορά των πόρων ε, γίνεται τώρα και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα θα διαβιβάσει τι επιλογέ για το πρόγραμμα εργασία που υποστηρίζεται από τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν αργότερα αυτή την εβδομάδα προ εξέταση. Αν η Κομισιόν υιοθετήσει το σχέδιο σχέδιο εργασία το Δεκέμβριο και κοινοποιήσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα ότι έχει θετηθεί το σχέδιο, ο Οργανισμό Άμυνα θα ξεκινήσει ε, τον διαγωνισμό και αυτό μπορεί να γίνει ήδη τον Ιανουάριο του 2016, την πρόσκληση υποβολή προτάσεων. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη τη βιομηχανία και τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, η αμυντική βιομηχανία είναι ουσιαστική για τη στρατηγική αστυνομία τη Ευρώπη και την ικανότητά τη να δράσει. Με του εταίρου, η ΔΕΗ και η Κομισιόν συνεργάζονται στενά για να ενεργοποιήσουν τα μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουν την αμυντική βιομηχανία. Το έργο του οργανισμού επικεντρώνεται στα εξή καταρχήν να διευκολύνει τη συμμετοχή 11 ε, μελών από την κεντρική, κρατών μελών από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη σε συνεργατικά προγράμματα. Ε, τώρα ολοκληρώνουμε μια χώρα ειδική για τις χώρες αυτές και τις βοηθούμε να ξεπεράσουν τα εμπόδια για την αμυντική συνεργασία ε, εντός της βιομηχανικής και τεχνολογικής αμυντικής βάσης. Συγκεκριμένες προτάσεις θα κατατεθούν για συζήτηση το πρώτο μισό του επόμενου έτους η εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για την ε, αλυσίδα εφοδιασμού και ένα σχέδιο δράση για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, προκειμένου να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στι αγορέ εφοδιασμού, ευκαιρίε επιχειρηματικέ, πληροφορίε για την αγορά και χρηματοοικονομικά. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση τη Ένωση ε, μέσω τη ε, αλληλεπίδραση με την Κομισιόν. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα έχει εντοπίσει πηγέ άμυνα για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει και ομοδοποιήσει όπω το κόσμο, το ΕΣΥΦ και η συνεργασία και η συνεργασία εταιρική σχέση με ε, το Enterprise Europe Network. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει πέντε εργαστήρια στα κράτη-μέλη το 2015 και σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε ακόμη τέσσερα το 2016. Επίσης, ε, ασφάλεια του εφοδιασμού προκειμένου να προωθήσουμε περαιτέρω την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία πολιτική υποστήριξη μεταξύ των κρατών μελών. Ο οργανισμός συνεχίζει να επιδιώκει διακυβερνητικές δράσεις που εγκρίθηκαν από τους υπουργούς το Μάιο του 2015 ως συνεισφορά στον οδικό χάρτη της Κομισιόν για να έχουμε ένα ευρύ καθεστώς εφοδιασμού. Ο οργανισμό θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν για να αναπτύξουν τι τελικέ προτάσει για τον οδικό χάρτη. Προτάσει ορισμένων κρατών μελών να ενδυναμώσουν περισσότερο την ασφάλεια του εφοδιασμού επίση αναλύονται. Παραδείγματο χάρη, μια πιθανή απόφαση του Συμβουλίου για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Σε σχέση με τις ευρύτερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικεντρωθώ στον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό, στο ΣΕΖΑΡ, στο ΡΙΤΣ και την ενέργεια. Ε, το ΣΕΖΑΡ και ο νέος Ευρωπαϊκός ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνος διευκολύνει το συντονισμό των ε, θεατρικών απόψεων, ο τρόπος, οι τρόποι ανάπτυξης του, Ευρωπαίου, του ευρωπαϊκού ουρανού μαζί με ΝΑΤΟ εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015. Συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ε, ενός Συμβουλίου ε, Στρατιωτικού Συμβουλίου για την Αεροπλοεία που θα προβαίνει σε συντονισμό και συνεργασία με τα κράτη και του διεθνεί οργανισμού, προκειμένου να μην υπάρχουν αρνητικέ συνέπειε σε εθνικέ και συλλογικέ, αμυντικέ ικανότητε. Οι προτεραιότητε του Οργανισμού Άμυνα είναι να διασφαλίσει τι ε, επιχειρησιακέ ε, ανάγκε ε, στο ΣΕΣ, στον Ευρωπαϊκό Ουρανό, Επίσης, να διευκολύνει τη στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα, τους οργανισμούς και τον ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεννόησης με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης του ΣΕΣΑΡ τον Ιούνιο του 2015 και εκεί εντοπίζονται στρατιωτικά project και προετοιμάζονται ε, προτάσεις για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τις προσπάθειες που γίνονται από τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσει κούσια σύμμορφωση των στρατιωτικών συστημάτων με τους κανονισμού ε, του Ευρωπαϊκού Ουρανού. Ε, πάντοτε τονίζαμε το ότι πρέπει οι στρατιωτικέ δυνάμεις να έχουν πρόσβαση στον ενέργειο χώρο για σκοπούς ε, ε και άμυνας. Οι, οι θα θα υποβληθούν στο ΙΝΕΑ που θα λήξει το Φεβρουάριο του 2016. Αυτά τα 42 project ε, καλύπτουν συστήματα εδάφους μέχρι πλατφόρμες ενέργειας και επίσης συγκεκριμένε μελέτες. Τώρα για το REACH. Ο κώδικας δεντολογίας για τις εξαιρέσεις άμυνας του ΙΤΣ που υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη το Μάρτιο του 2015 είναι ένα μεγάλο βήμα προς την εναρμόνιση των εθνικών διαδικασιών στο να χορηγήσουμε εξαιρέσει άμυνα στο ΡΙΤΣ, ο στόχο είναι να μειωθεί το κόστο και η γραφειοκρατία. Ε, μαζί με τα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με την Κομισιόν και ε, την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, προετοιμάζουμε έναν οδικό χάρτη για να διευκολύνουμε το συντονισμένη δράση, προκειμένου να εντοπίσουμε και να επικεντρώσουμε τι προσπάθειε για να μειώσουμε τον αντίκτυπο του ΡΙΤΣ στην άμυνα ενώ συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Αυτός ο χάρτης πορείας ε, θα πρέπει να ετοιμαστεί το πρώτο εξάμεινο του 2016. Επίση, έχοντα κατά νου το ενδιαφέρον των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μενών, όπω το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνα, ε, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα μπορεί να παίξει συντονιστικό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι απόψει τη κοινότητα στρατιωτική συνολικά συντονίζονται και στέλνονται στην Κομισιόν και στον Οργανισμό Χημικών. Την ενέργεια. Η χρήση ενέργειας ε, στο στρατό δεν αφορά μόνο την αύξηση της αντοχής. Το να αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα για την ανάπτυξη των μέσων είναι κάτι ουσιαστικό, όπως και να έχουμε μια κατανόηση ότι η χρήση της ενέργειας στις εγχώριες επιχειρήσεις μας είναι εξίσου σημαντική. Ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας οργανώνει το φόρουμ διαβούλευσης εκ μέρους της ΓΔΕ με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για βιώσιμη ενέργεια στον τομέα άμυνα και ασφάλεια. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στι 14 και 15 Ιανουαρίου. Ο στόχο αυτή τη διαβούλευση είναι να εξετάσει την εφιστάμενη ενεργειακή νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιολογήσει πώ εφαρμόζεται στο ε, στρατιωτικό τομέα να διευκολύνει και υποστηρίξει project που θα προωθήσουν την αποτελεσματικότητα την ενεργειακή στο στρατιωτικό τομέα, να εξετάσει τις εφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και να εντοπίσει νέους μηχανισμούς που είναι κατάλληλοι για το στρατιωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα συνεισφέρουν στο ε, να έχουμε καλύτερους ενεργειακούς στόχους. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό η διαβούλευση αυτή να καταλήξει στην ανάπτυξη συστάσεων εκ μέρους του τομέα άμυνας για να διευκολύνει την πρόοδο. Ο μελλοντικό ρόλος και κατεύθυνση του οργανισμού επίσης ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των Υπουργών στις 17 Νοεμβρίου. Δεδομένη τη σημερινή κατάσταση ασφαλεία, έχουμε πέντε τομεί όπου πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμενας. Καταρχήν, το σχέδιο ανάπτυξη ικανοτήτων που αναπτύχθηκε από του εμπειρογνώμονε των κρατών μελών και αντικατοπτρίζει τι απαιτήσει του πρέπει να μεταφραστεί σε δράσει. Οι ειδικοί χάρτε για μελλοντικά συνεργατικά project επίση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ω ένα πραγματικό μέσο για αμυντικό σχεδιασμό και για την υποστήριξη τη περιφερειακή συνεργασία και άλλων πρωτοβουλειών όπως ε, το πλαίσιο της έννοιας των δεύτερων. Έχουμε την εξαίρεση από το ΦΠΑ, ένα πιθανό ταμείο για την άμυνα, τυποποίηση και πιστοποίηση και η σύνδεση της άμυνας με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Τρίτον, όπως γνωρίζετε, οι περικοπές ε, στην ε, άμυνα έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων και σε διάφορες προκλήσεις ε, στον τομέα της ασφάλειας, στην προπορισκευαστική δράση θα έπρεπε να είναι ο καταλήτης για μεγαλύτερη δέσμευση στην έρευνα και τεχνολογία στην άμυνα και να οδηγήσει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που θα συμπεριληφθεί στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα αντιμετωπίσει τις μελλοντικέ προτεραιότητες ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέταρτον συστηματικές ε, συνέργειε μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού τομέα, χρησιμοποιώντα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα ω διαπαφή. Χωρί να θίγεται η εθνική κυριαρχία, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τι ε, τις ευκαιρίες ε, που προσφέρονται από τι συνέργειε αυτέ, παραδείγματος χάρη σε τομεί, όπω ε, η θαλάσσια ασφάλεια, η ενέργεια και το περιβάλλον, το διάστημα και ο νέος Ευρωπαϊκό Ουρανό. Και τέλο, οι ευκαιρίες που προσφέρονται από την χρηματοδότηση της Ένωσης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι σε θέση να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών. Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης της Κομισιόν. Αυτό θα γίνει μέσω άμεσης δέσμευση στη διαδικασία και στη συνέχιση του έργου μας σε κύριους τομείς όπως είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού, μικρές και μεσές επιχειρήσεις και η προπαρασκευαστική δράση. Αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια ισχυρή ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη η αμυντική βιομηχανία που θα υποστηρίζει τι ανάγκε μα οι ικανότητε Πριν να κλείσω πρέπει να πω και κάτι τελευταίο, τον προπολογισμό. Όπω ε, όλοι μπορεί να γνωρίζετε, αντιμετωπίζουμε για το 2016 και για έκτο χρόνο στη σειρά έναν ε, προπολογισμό που παραμένει σταθερό. Τώρα αντιμετωπίζουμε το παράδοξο ενό προπολογισμού που μειώνεται περισσότερο σε πραγματικού όρου, ενώ έχουμε όλο ένα και περισσότερα καθήκοντα. Αυτό θα σημαίνει ότι κάποιε από τι δραστηριότητε του πλαισίου μα του τριετού θα αναβληθούν, θα μειωθούν σε κλίμακα ή θα καταργηθούν εντελώ. Είμαστε λοιπόν σε μια κρίσιμη συγκυρία. Αν κάνουμε σωστά τα πράγματα, μπορούμε να διασφαλίσουμε στρατηγική αυτονομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να έχει ρόλο ως πάροχος ασφαλείας και ως αξιόλογος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Αλλά πρέπει να δράσουμε τώρα και θα πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα μέσα, τους κατάλληλους πόρους. Σας ευχαριστώ. thank Σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ. Ήσασταν ιδιαίτερα αναλυτικός ε, και συνολικός, όμως είμαι σίγουρος, ε, σίγουρη ότι υπάρχουν ακόμα ερωτήματα. Κύριος Γκάλλαρ θα ήθελα να μιλήσει. Ναι, σας ευχαριστώ ε, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, συλλογική απεικόνηση. Ε, έχουμε τα έγγραφα στην μπροστά μας Ναι, αυτό το οποίο έχουμε δει ε, συνήθως ε, τα τελευταία έξι χρόνια ε, και παραμένει σταθερό και οφείλεται στη Βρετανική κυβέρνηση. Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Δυστυχώς έτσι είναι. Η δική σας κυβέρνηση δυστυχώς μπλοκάρει μία αύξηση και με, ενώ ταυτόχρονα οι προκλήσεις και οι απειλές γίνονται όλο και περισσότερες. Ε, γι' αυτό το λόγο ας ε, κατονομάσουμε και ας δείξουμε το δάχτυλο, δεν, ε, ας τονίσουμε ποιοι ευθύνονται. Ε, θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε με αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν και θα πρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες δράσεις, όμως δεν είναι αυτό το βασικό αυτή τη στιγμή. Είχα ένα ε, γεύμα σήμερα ε, μαζί με έναν εκπρόσωπο της Βρετανικής Βιομηχανίας και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, διότι η αγορά τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους απασχολεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Και γι' αυτό το λόγο ίσως θα πρέπει να ασκήσουν και την αναγκαία πίεση προς την κυβέρνησή τους, ούτως ώστε να υπάρξει ροή των αναγκαίων ε, πόρων ήμουν μεταξύ αυτών που ξεκίνησαν το πιλωτικό πρόγραμμα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας μαζί με την ε, κοινή ε, προσπάθεια ε, οδήγησε ούτως ώστε στις 17 Νοεμβρίου να υπογραφεί αυτό και να δούμε χρήματα στον προϋπολογισμό. Προσθέσατε επιπλέον δεν θα επιστρέψω σε όλες τις λεπτομέρειες, όμως ένα επιπλέον θέμα στο οποίο αναφερθήκατε 32 συνολικά προγράμματα για το ΣΥΖΑ για το ΣΥΖΑΡ από πού θα προέλθουν τα συγκεκριμένα ε, κονδύλια και τα 28 κράτη-μέλη, ε, αυτά τα οποία έχουν ε, αεροπορικές δυνάμεις, θα παράσχουν τα μέσα ούτω ώστε ε, να μπορούν να πετάνε στο ε, European Single Sky. Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω. Αλλιώς άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία ταυτοποιήθηκαν ε, ήδη από το Δεκέμβριο του 2013 ήταν, αφορούν την κυβερνοάμυνα καθώς επίσης και τα drones και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε και γι' αυτό το λόγο ε, και αυτά αποτελούν ε, ένα λόγο για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Θα έχετε λοιπόν την πλήρη υποστήριξη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να μπορέσετε να κάνετε όσα χρειάζονται. Σας ευχαριστώ. Κύριε ε, Πρέσβη μέκ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ε, πράγματι είστε ένας ε, πάρα πολύ καλός εκπρόσωπος ε, του έργου σας. Ε, αν γνώριζα ποιος είναι ο ανώτερός σας, αν υπάρχει η κυρία Μογερίνη, τότε την επόμενη φορά που θα τη δω θα της πω ότι είστε ένας άριστος διευθυντής. Αυτό όμως δεν σημαίνει βέβαια ότι συμφωνώ με, τα, ε, όλα όσα έχετε αναφέρει. Έχω μπερδευτεί λιγάκι σχετικά ε, με ε, όσα είπατε στο, στα σχόλιά σας. θα σας παραφράσω τώρα λίγο αν ε, κάνω κάποια λάθη τότε, ε, ε, τότε διορθώστε με. Χρειαζόμαστε πραγματικά γεγονότα σαν αυτά στο Παρίσι και ό,τι συνέβη στις Βρυξέλλες, ούτως ώστε να αναλογιστούμε έναν στρατό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι τέτοιο νομίζω είπατε. Και δεν ξέρω, όταν έρχεται από κάποιον, ε, από την ειρηνική χώρα, την Αυστρία, ε, ο στρατός ε, και ουδέτερη Αυστρία, ξέχασα να αναφέρω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήξερα ότι θα γελάσετε. Οι Γερμανοί πάντοτε γελάνε όσον αφορά τους Αυστριακούς. Αν λοιπόν η σωστή απάντηση σε αυτό το οποίο αναφέρατε είναι όντως η στρατιωτική απάντηση, τουλάχιστον από ε, το μέρος όπου μεγάλωσα εγώ, και ευτυχώς ε, δεν υπήρχαν εκεί τέτοια περιστατικά, όμως η σωστή απάντηση, όπως έμαθα εγώ τουλάχιστον, είναι η αστυνομία, το δικαστικό σύστημα, και ίσως ε, οι μυστικές υπηρεσίες ε, για να ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα, αν είναι αυτή η σωστή λέξη. Και όχι ο στρατός. Ναι, στους δρόμους στο Παρίσι αλλά και στις Βρυξέλλες βλέπω στρατιωτικό προσωπικό. Κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο στην Αυστρία. δεν επιχειρηματολογώ για αυτό τον κοινό ευρωπαϊκό στρατό που οροματίζεστε και ίσως να είναι αναγκαίος για να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από την ε, απαλή δύναμη την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον. Όμως ε, το να αναφέρουμε αυτά τα γεγονότα, τα τρομακτικά γεγονότα σε Βρυξέλλες και Παρίσι και να τα χρησιμοποιούμε ε, για να ως ευκαιρία για την εφαρμογή της ε, ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πάλι όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το, ε, δεν το χρειαζόμαστε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Όμως από την άλλη όταν το σκέφτομαι πάντοτε θα μας συγκρίνουν με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη. Αν αρχίσουμε λοιπόν ε, να δημιουργούμε μια ευρωπαϊκή άμυνα, ένα τέτοιο σύστημα, τότε θα μας συγκρίνουν με τους Αμερικανούς, με τους Ρώσους, με τους Κινέζους Και αναρωτιέμαι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε ένα τέτοιο επίπεδο, το επίπεδο των Αμερικανών. Ξέρετε πόσα δαπανούν για τον στρατό τους ακόμα και σε σχέση με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Θα μπορέσουμε λοιπόν ποτέ να φτάσουμε ένα τέτοιο επίπεδο. Δεν είμαι βέβαιος και δεν ξέρω αν θα ήταν μια καλή ιδέα. Σας ευχαριστώ κύριος ε, Κάμπλ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αναφέρατε ε, την πρόθεση μιας ενιαίας ε, βιομηχανίας ε, άμυνας και την εφαρμογή αυτή σε όλη την Ευρώπη, όμως χωρίς να υπάρξει μια αύξηση του προϋπολογισμού, η Μεγάλη Βρετανία να κρατάει το 2% του ΟΕΠ σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, Πώς λοιπόν ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι ωφέλιμο ναι. ιδιαίτερος για την ε, Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι οι χώρες που δαπανούν τα περισσότερα όσον αφορά την άμυνα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πάτμαντς. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Κύριε Πρέσβη, θα περιμένουμε να βάλετε ακουστικά excuses later was. Ζήτω συγγνώμη που ήρθα κάπως καθυστερημένη. Είχα κάνει κάποιο προπαρασκευαστικό έργο, αλλά ε, ήρθα στο τέλος της παρουσίασής σας. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και το ανέφεραν και άλλοι ομιλητές είναι τι θα κάνουμε μετά το Παρίσι. Νομίζω ότι αν ε, κάποιο εργάζεται στο Κοινοβούλιο, πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, έρχεται εδώ, το πρώτο που μα απασχολεί, πρώτο μα μέλημα είναι τι θα κάνουμε μετά το Παρίσι. Εσείς συναντηθήκατε στις 17 Νοεμβρίου, μερικές μέρες μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και πραγματικά θα ήθελα να ξέρω πώς επηρέασε το Παρίσι τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε εσείς σήμερα. Ελπίζω ότι το Παρίσι άνοιξε κάποιον τα μάτια. Ε, άρχισαν κάποιοι να κατευθύνονται σε κάποιο διαφορετική κατεύθυνση. Κάποιοι είπαν ότι δεν νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά εγώ νομίζω ότι ε, θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Εάν μετά από το Παρίσι δεν μας έχει πείσει ότι χρειαζόμαστε κάποια κοινή άμυνα, έναν ευρωπαϊκό οργανισμό άμυνα, τότε τι άλλο πρέπει να συμβεί για να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και να ασχοληθούμε με αυτό. Και κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για το εξή. Ε, καλέσατε τον ε, καθηγητή Μάτελαρ, ο οποίος θα έρθει αργότερα και θα μας εξηγήσει λίγο ε, ποιε είναι οι συνέπειε της επίκλησης του άρθρου 42 παράγραφος 7 και επειδή ακριβώς ξεκίνησε αυτό να δούμε και τι συνέπειες θα υπάρχουν. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα να σας ζητήσω είναι ότι ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή άμυνα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι άλλαξε το Παρίσι στο πρόγραμμά σα. μου απαντήσετε τίποτα θα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Οπότε ελπίζω ότι τουλάχιστον το Παρίσι έχει προκαλέσει κάποιε αλλαγέ. Και δεύτερον, ε, από ό,τι έμαθα, ο προπολογισμό έχει παγώσει. Ποια είναι τα κριτήρια για να σταματήσουν οι εξελίξει εκεί. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστώ για τι απαντήσει. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για το λόγο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς ε, για την αναλυτική παρουσίαση. Εγώ προσωπικά κατάγομαι από το Μόναχο και όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε κοντά στην Αυστρία και δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη που και εγώ αντιπροσωπεύω τις ίδιες απόψεις όπως και ο φίλος μου από εδώ. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα επίσης Ιδιαίτερος λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω ότι ο διαχωρισμός των στρατιωτικών ε, δράσεων και πολιτικών δράσεων από την πλευρά της αστυνομίας για παράδειγμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερος ε, λαμβάνοντας υπόψη μας τα όσα έχουν συμβεί στο Παρίσι θα ήθελα να σας καλέσω να μην συγχαίουμε αυτά τα πράγματα. Επίσης ε, μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι στον το στρατιωτικό τομέα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ε, δαπάνες και γι' αυτό το λόγο η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, θα... Θα ήθελα να είμαι λίγο επιφανειακός, ε, δεν είναι όμως αναγκαίο να συνεχίσουμε έτσι όπως το κάνουμε τώρα. Θα ήθελα επίσης να, ένα συγκεκριμένο, να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Αναφερθήκατε στα drones όπως γνωρίζετε η Γερμανία, η χώρα μου, ασχολείται ιδιαίτερος ε, με αυτό το θέμα, οπότε θα μπορούσατε να αναλύσετε το συγκεκριμένο θέμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε έτσι ε, η διαδικασία των ερωτήσεων και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ντόμεκ ε, να δώσει απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για τις παρεμβάσεις σας και για τα καλά λόγια που είπατε για το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και τώρα θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Καταρχάς, προς τον κύριο Γκάλερ και τα 32 προγράμματα τα οποία επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη προκειμένου να τα υποβάλουμε ε, στην πρόσκληση ναι, για την συγχρηματοδότηση. Όπως γνωρίζετε, ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός είναι ένας από τους τομείους ε, στους οποίους επικεντρώνεται ιδιαίτερα ο οργανισμός μας, διότι είναι μεγάλη ανησυχία για τους επικεφαλείς ε, των αεροπορικών δυνάμεων. Πρέπει να το καταφέρουμε αυτό. Ξέρετε πριν από κάποια χρόνια ότι υπήρχε ανησυχία ότι η πολιτική αυτή γινόταν ε, απόλυτα απομονωμένη χωρίς ε, να λαμβάνουμε υπόψη και τι συνέπειες μπορεί να υπάρχουν και για το στρατό μας. Την Άνοιξη, όταν έφτασα εγώ στον οργανισμό και εξετάζαμε τα διάφορα στοιχεία που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Ρωνό, εξετάζαμε πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα Υπουργεία Άμυνας ε, να προετοιμάσουν τις προσκλήσεις ε, της υποβολής των προσφορών για αυτό το διαγωνισμό και ε, να δούνε και τι γίνεται με τον εναόριο χώρο τους. Επειδή πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκτελεστεί για πάνω από 30 χρόνια, θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε κάποια προγράμματα, ένα-δυο, τα οποία θα πρέπει να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να έχουν υποβληθεί αυτές οι προτάσεις και αν το καταφέρουμε αυτό θα αποτελεί επιτυχία, διότι... Ε, ο μηχανισμός του Υπουργείων Άμυνα δεν είναι προετοιμασμένος για να δραστηριοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό το οποίο μας εξέπληξε όταν τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και είχαμε αρχικώς 97 ε, δηλώσεις προθέσεων, έγινε ένα έλεγχο με τα κράτη-μέλη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα ε, επιλέξουμε αυτά τα οποία είναι ε, τα πιο πολλά υποσχόμενα και αυτά τα οποία απαιτούνται περισσότερο και τώρα τα προετοιμάζουμε από τεχνική σκοπιά και θα ξεκινήσουν να ολοποιούνται. Ε, θα υπάρξει υποβολή για χρηματοδότηση, θα πρέπει να γίνουν πολλές προσαρμογές στα συστήματα ATM στις επίγειες βάσεις, λόγω μάλλον των συστήματων ATM και επίσης και με το ε, μεταφορικό στόλο. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές ούτως ή άλλως προβλέπονταν σε εθνικό επίπεδο Επομένως τώρα θα μπορέσουν ε, τρόπον την να αποζημιωθούν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ε, τα σχέδια οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να είναι αντίστοιχα της χρηματοδότηση. Αυτό λοιπόν για αυτό το οποίο με ρωτήσατε έχω να πω απάντηση. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Φρόιντ, ε, Ε, για το τι εννοούσα με αυτή την αφύπνιση. Και είπατε ότι αμφιβάλλεται αν η σωστή απάντηση είναι ο στρατός. Νομίζω ότι όπως έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, δεν μπορούμε πλέον να αναφερόμαστε στην ασφάλεια η οποία σταματά στα σύνορα. πού σταματάει το πολιτικό και πού αρχίζει το στρατιωτικό σκέλος στην αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν γνωρίζουμε. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω ότι αυτό θα συμβαίνει και στις μελλοντικέ κρίσεις, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές τις συνέργειες πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους. Και δεδομένης και της ε, αρμοδιότητας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτουμε όλες τις πτυχές που αφορούν τον υβριδικό πόλεμο. Αυτό σημαίνει υβριδικός πόλεμος. Σημαίνει ότι υπάρχει εισρωή από πηγές οι οποίες δεν είναι αμυγός στρατιωτικές, αλλά μπορούν να γίνουν αν θέλουν να απαντήσουν σε μία απειλή σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, είπατε ότι αυτό αφορά περισσότερο την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Ε, αμφιβάλλω ότι είναι αυτή η σωστή απάντηση, διότι η απάντηση όπως θα δούμε από το άρθρο 42.7 ε, θα είναι κάτι το οποίο θα καλύπτει και ένα πιο σκληρό σκέλος και γι' αυτό άλλωστε έγινε και επίκληση του άρθρου αυτού. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία και όχι μόνο αυτά τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με συντονισμένο τρόπο. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε. Πριν από κάποια χρόνια ε, ελάχιστοι θα ήταν ε, ε, διατεθειμένοι να συζητήσουν θέματα του στρατού και συμμετοχή σε δραστηριότητες εποπτείας εντός της χώρας μας. Κάποιοι μάλιστα θα ήταν και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Αλλά δεν νομίζω ότι οι πολίτες σήμερα, οι οποίοι χρήζουν προστασίας, θα είναι τόσο αντίθετοι. Έχει γίνει λοιπόν αυτό το κβαντικό άλμα στο πώς εξετάζουμε εμείς οι ίδιοι την ασφάλεια. Και αυτό είναι με δύο λόγια. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε απλά πλέον ως αμυγός στρατιωτική ή με αμυγός πολιτική απάντηση. η ε, υπόλοιπη παρέμβασή σας για τη σύγκριση με άλλες μεγάλες δυνάμεις ε, και το πώς μπορούμε να φτάσουμε στο ύψος τους, αν μπορούμε να φτάσουμε στο ύψος τους, θα πρέπει ίσως να φτάσουμε στο ύψος τους, ε, Εμείς εδώ εργαζόμαστε για την παγκόσμια στρατηγική και θα πρέπει να έχουμε ένα έγγραφο τον Ιούνιο το οποίο θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον ως Ευρωπαίοι. Και από εκεί θα πρέπει να δούμε τι ρόλο θέλουμε να διαδραματίσει και το στρατιωτικό στοιχείο. θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να, βλέπε, ε, να, να εξετάζεται ως κάτι απομονωμένο, αλλά ως τμήμα των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, θεωρώ ότι υπάρχει κάποια εξίσωση ε, βάσει της οποίας εάν κάποιος θέλει να είναι παγκόσμιος παράγων που μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα ε, χωρίς εμείς να δώσουμε τη δέουσα σημασία και στη στρατιωτική πτυχή δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε παγκόσμιοι παράγοντες και ε, να παρέχουμε ασφάλεια με οποιονδήποτε τρόπο εάν δεν υπάρχει και μία ραχοκοκαλιά στρατιωτική. Για την ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία και την κατεύθυνση αυτή προς μία ενιαία αγορά με τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν για κάποια κράτη-μέλη τα οποία έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη βιομηχανία. Ε, η αλήθεια εδώ είναι και το τι ε, κίνδυνο ελοχεύει για τις διάφορες θέσεις εργασίας άμα ανοίξει η αλυσίδα εφοδιασμού ε, είναι ότι οι συνέπειες θα υπάρχουν ακόμα και για τις μεγάλες βιομηχανίες. Δεν θα επιβεώσουμε μακροπρόθεσμα εάν έχουμε το, τέτοια κοντόφθαλμη οπτική. Παραδείγματο χάρη, στον τομέα των πυράβλων υπάρχει μια επιχείρηση η οποία ε, είναι στην πρώτη γραμμή, η NBDI, η οποία ε, συστήθηκε ε, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα συστήματα των κρατών μελών και συμπεριλαμβάνοντας τα όλα. Μόνο έτσι κατάφερε να μείνει ανταγωνιστικό και στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό ακριβώς ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι αμυντικές μας βιομηχανίες είναι να επιβιώσουν είναι η συνεργασία στην άμυνα. Δεν πρόκειται για δυνατότητα επιλογής. Εάν θέλουμε να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία, τα προγράμματα τα οποία ξεκινούν σε εθνικό επίπεδο, πολύ εύκολα θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι βιώσιμα από οικονομική σκοπιά. Και επίση, αν κάποιο θέλει πραγματικά να υπάρχει συνεργασία στην άμυνα, τότε τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει ε, να θέλουν να έχουν πρόσβαση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους και φυσικά αυτό θα πρέπει να γίνει με κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα οργανώσουμε εμείς όλα όσα πρέπει να κάνει η αγορά, αλλά θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τον κλάδο για το τι αγορά θέλουμε να αναπτύξουμε σε συνεργασία. Εάν δεν γίνει αυτό, ακόμα και οι μεγάλες ε, χώρες μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ε, θα καταλήξουν χωρίς βιομηχανία. Αυτό είναι σαφές και ξεχάστε αυτές τις μικροπολιτικές ε, των θέσεων εργασίας, ε, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμα τα πράγματα, διότι βραχυπρόθεσμα, τώρα που βλέπουμε να δαπανώνται περισσότερα ε, στην άμυνα, στους προπολογισμούς σε κάθε χώρα. Εάν ξοδέψουμε και σπαταλήσουμε χρήματα θα πάνε χαμένα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν μεγαλύτερε επενδύσεις στην άμυνα, αλλά καλύτερες επενδύσεις στην άμυνα. Και καλύτερε επενδύσεις σημαίνει συνεργασία στην άμυνα. Για την ερώτηση της κυρίας Βόντεμ. ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δεν έχει επιχειρησιακό ρόλο. Επομένως η απάντηση δική μας είναι διαφορετική φύσεως. Τα γεγονότα στο Παρίσι επεσήμαναν αυτό που έλεγα και στον κύριο Φρόιντ, ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι συνεργασίας ε, πολιτικής στρατιωτικής πτυχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε στο μέλλον. δύσκολα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις που θα περιλαμβάνουν σαφώς μόνο στρατιωτική προσέγγιση. Θα πρέπει να είναι ένα αμάλγαμα διαφόρων στοιχείων που θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Τώρα, ελπίζω ότι όπως είπαν και οι υπουργοί σας ε, στην ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, άμυνας ε, ότι αυτό θα είναι η αφύπνιση που χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια αμυντική Ευρώπη. Όσον αφορά το προϋπολογισμό ε, που έχει παγώσει, που σημαίνει ότι τα τελευταία έξι χρόνια χάθηκε πάνω από το 12% του επιχειρησιακού προϋπολογισμού και κυρίως αυτό πλήττεται. Ε, είχαμε μια αύξηση 10% που μπλοκαρίστηκε λόγω βέτο και αυτό ήταν να αφιερωθεί όλο τον επιχειρησιακό ε, ε, προϋπολογισμό και ένα πολύ μικρό ποσοστό θα διατεθεί στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό από το 97% αυτό που δίνουμε. το συζητούσα τώρα με τα κράτη-μέλη για το πώς μπορούμε να ε, αυξήσουμε τις δραστηριότητες μας, γιατί πρέπει κάπως να τις αυξήσουμε ή θα πρέπει να καθυστερήσουν κάποια προγράμματα. Ένα στοιχείο το οποίο καταφέραμε με τη νέα απόφαση του Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου είναι ότι μπορεί να λάβει περαιτέρω έσοδα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, ε, άμυνας. Ε, το πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Γκάλερ είναι μια κλασική περίπτωση που μπορεί να προέρχεται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αλλά μπορούμε να λάβουμε και επιπλέον προϋπολογισμό σε εθελουσία βάση από τα κράτη-μέλη. Έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη βοήθεια. Ε, δεν φαίνονται και πολύ άσχημα τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν θα λάβουμε αυτό το ποσό που θέλουμε. δεν μου αρέσει και αυτός ο ad hoc τρόπος να ζητούμε χρήματα και ενώ όταν εμείς άπρεπε να μπορούμε να έχουμε πόρους και όχι να παίζουμε με τα νούμερα. Ζήτησε επίσης ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινους πόρους, γιατί είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε και ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε ένα μικρός οργανισμός, 120 εμπειρογνώμονες και αν εγώ ε, έχω κάποιους περαιτέρω εμπειρογνώμονες, τότε θα μπορέσω να προχωρήσω. Τέλος, Κύριε Μπούχνερ, για το ΑΡΠΑΘ. Πέραν του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν τα τέσσερα κράτη-μέλη για αυτή τη μελέτη του ορισμού και η χώρα σας και άλλες τρεις, Εμείς ε, θα επικεντρωθούμε κυρίως ε, πρώτον να διασφαλίσουμε ότι τα στρατιωτικά drones μπορούν να ενταχθούν εύκολα στον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο. Γιατί ξέρετε ότι αυτό ε, ήταν πρόβλημα στο παρελθόν και χρειάζεται και μία διπλή στρατηγική διπλής χρήσης για τις πτυχές ασφαλείας και αυτό μας ανέθεσαν να προωθήσουμε οι Υπουργοί. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πτυχές του αξιόπλου, το οποίο ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όλα όσα έχουμε κάνει στον οργανισμό όσον αφορά την ε, ε, ευρωπαϊκή στρατηγική ε, ως προς το αξιόπλο και τη δυνατότητα των προδιαγραφών είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουμε φροντίσει να υπάρχει βοήθεια και από τα κράτη-μέλη ώστε να μην χάσουμε ούτε από οικονομική σκοπιά αλλά ούτε και χρόνο. Και τέλος, το βασικό πρόγραμμα του ΑΡΠΑΣ, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, Θέλουμε να παραμείνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό θέλει να διασφαλίσει ο οργανισμός μας, το οποίο αργότερα θα ε, είναι ανοιχτό για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που θέλουν να συμμετέχουν. Δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτό το στρατηγικό μέσο, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της αγοράς των drones ε, σε 10 χρόνια, και το τι θα ε, αντιπροσωπεύει αυτό για τον κλάδο, αλλά και γιατί θεωρώ ότι θα είναι από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους ε, ε, η βιομηχανία των εναέριων μεταφορών θα μπορέσει να αναπτύξει δεξιότητες τις οποίες τώρα αφιερώνουν σε εναέριες μάχες. Ξέρετε ότι η επόμενη γενεά δεν προβλέπεται προς το παρόν, αλλά ε, υπάρχει μια πολύ σημαντική ομάδα μηχανικών ε, με γνώσεις και δεξιότητες που αν τους αφήσουμε να διαλυθούν ε, θα είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια να τους ε, ξανασυγκεντρώσουμε και να ξεκινήσουν τα πράγματα από την αρχή. Πρέπει κάπως να καταφέρουμε να διατηρήσουμε αυτές τις στρατηγικές δυνατότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρέσβη Τομέκ για αυτή την ε, πλήρη ενημέρωση και για τις εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις σας. Είχαμε μία πλήρη ενημέρωση για την ε, συνεδρίαση του Υπουργικού Διευθυντικού Συμβουλίου. Επίσης σας ε, ευχαριστούμε που απαντήσατε και στις ερωτήσεις. Βασιζόμαστε στο να επανέλθετε εδώ ενώπιον της Επιτροπής μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσω τώρα το επόμενο σημείο τη ημερική διάταξη. Παραμείνετε παρακαλώ στην αίθουσα. Okay. Gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Είναι τιμή μου να καλωσορίσω τον ε, καθηγητή Ρόντερικ Πάρξ, ο οποίος είναι ανώτερος αναλυτής του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας. Κύριε Πάρξ, Κύριο Πάρξ θα κάνει μια συζήτηση μαζί μας ε, για το θέμα της παράνομης διακίνησης μεταναστών και τις συνέπειες αυτής για την εξωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλο τον αντίκτυπο στην ασφάλεια του θέματος της παρανομής διακίνησης ε, μεταναστών. Θα πρέπει να δούμε φυσικά και τι γίνεται στο Βρυτό, στη Βενησία. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και τα γεγονότα στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιες συνδέσμοι και έχουμε και συνέπειες και στην εσωτερική μας ασφάλεια και φυσικά δεν θα πρέπει να τα περιμερίσουμε τα ζητήματα αυτά. με ενημέρωσαν ότι είναι εδώ η εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κτίριο. Ίσως αργότερα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την απόψή σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Καταρχήν ο κύριος Πάρξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και την εισαγωγή θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για το πώς έχουν τα πράγματα, μέσα σε 15 λεπτά περίπου. Αλλά αν μπορώ να σας δώσω μια ιδέα σήμερα είναι ότι τα Δυτικά Βαλκάνια κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργική διάλυση Μπορεί να φαίνεται βαρετό όρο, αλλά το διάλεξα πολύ προσεκτικά. Για τα τελευταια 20-25 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δημιουργήσει λειτουργική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Η κλασική ιδέα ε, του να υπάρχει διασυνοριακή οικονομική συνεργασία προκειμένου να υπάρχει από ε, εθνικιστικών πολιτικών ε, αυτή όμως η διάλυση ε, έρχεται επειδή οι πιο αποτελεσματικοί οικονομικοί παίκτες στα Δυτικά Βαλκάνια αυτή τη στιγμή είναι οι διακινητές ανθρώπων και η παραοικονομία και και είναι πολύ αποτελεσματική στο να διακινούν, να διακινούν μεγάλο αριθμό ατόμων διασυνοριακά. Έτσι λοιπόν αυτό έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, οδηγεί σε πολιτικό και διακερματισμό και σε κοινωνικού χαρακτήρα διαιρέσεις. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρουμε σε αυτό τον όρο τον που αφορά την λειτουργική διάλυση. Λοιπόν, θα σας δώσω αρχικά κάποιο ιστορικό πώς έχει η κατάσταση στα Βαλκάνια σε σχέση με τη μετανάστευση και θα κάνω τρία σχόλια για να απεικονίσω την κοινωνική και πολιτική διαίρεση. Καταρχήν, για το ιστορικό, να σας δώσω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία και η Ελβετία φέτος ε, είδαν περίπου ναι, 1.700.000 νέες αιτήσει ασύλου. Η ευρύτατη πλειοψηφία είναι αιτήσει που κατατίσσονται πρώτη φορά και εκεί που θα περιμέναμε ουσιαστικά μείωση είδαμε αύξηση. Στην Ελλάδα το Νοέμβριο είδαμε να έρχονται άνθρωποι από την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό, βλέπουμε περίπου 600 άτομα έως 6.000 άτομα ημερησίως να καταφτάνουν. Βλέπουμε περίπου 3 με 4.000 άτομα να μετακινούνται στα Βαλκάνια. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει εκεί τεράστια συσσόρευση και μιλάμε για μεγάλο αριθμό ανθρώπων που μετακινούνται σε ένα μικρό χώρο μεταξύ της Ελλάδας ε, και των κρατών μελών. Είναι απελπισμένοι οι άνθρωποι, απελπίζονται. Βλέπουμε τις ε, ροές να επανέρχονται στην Ελλάδα, Ναι, οδοί διακίνησης, ε, ε, χαράσσονται από την Ελλάδα στην Αλβανία και λόγω της συνεργασίας με την Τουρκία έχουμε και ίσως ενδυνάμει νέες οδούς από την Τουρκία στη Ρουμανία. Αυτή είναι μια καθολική εικόνα αν θέλετε. Τώρα αν μιλήσουμε για τα Βαλκάνια είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για τη Δυτικά Βαλκάνια, οι χώρες αυτές ε, δεν ε, είναι μόνο χώρες διέλευσης, αλλά είναι και χώρες προέλευσης. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου τα Δυτικά Βαλκάνια σε μπλοκ ε, ήταν ο δεύτερος ουσιαστικά τόπος προέλευσης και βλέπουμε πολλούς να έρχονται από το Κόσοβο του κοσφοπαίδιο στην Ουγγαρία, στη συνέχεια μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί Αλβανοί. Ε, ουσιαστικά παίρνουν το αεροπλάνο απευθεία για τη Γερμανία και καταθέτουν έτσι ασύλου αβάσιμε στι περισσότερε περιπτώσει. Και να σα πω συντομία πώ απάντησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η κύρια πρωτοβουλία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει hot spot στα σύνορα στα εξωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η υποδοχή, να γίνει διαλογή των ανθρώπων που ίσως θα μπορούσαν να επανακατασταθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εντοπιστούν και τα δίκτυα των διακινητών και να υπάρξει και λήψη πληροφοριών από τους ανθρώπους που είναι αντικείμενο εκμετάλλευση των διακινητών. Επίσης, χρησιμοποιούμε μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ε, πείσαμε τη Σερβία και τη Μακεδονία να το χρησιμοποιήσει για να μπορέσουν να οικοδομήσουν και αυτοί οι ικανότητες να υποδεχτούν τους μετανάστες το χειμώνα. Και επίσης ε, καθώς τα Δυτικά βουλκάνια είναι χώρες προέλευσης, ε, έχουν ε, θεσπιστεί μηχανισμοί εντός του προγράμματος απελευθέρωσης θεωρήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Και υπάρχει και μια συζήτηση για το αν μπορούμε να θεωρήσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια ως ασφαλείς χώρες προέλευσης αν κατατίθεται τη συλλου από υπηκόους των Δυτικών Βαλκανίων, μπορούμε να τους θεωρήσουμε ότι ε, ουσιαστικά είναι αβάσιμες αυτές οι αιτήσει. Αυτό είναι ουσιαστικά το ιστορικό. Τώρα, τρία σύντομα σχόλια, αν μου επιτρέπετε, για τα γεγονότα και το φαινόμενο της διακίνησης των ανθρώπων στα Βαλκάνια. Καταρχήν να πω ότι είναι πιο ευφυείς, πιο έξυπνοι διακίνητες από εμάς. Το Σεπτέμβριο η Γεροπόλη είπε ότι ίσως 30.000 άνθρωποι να εμπλέκονται στη διακίνηση και στην εμπορία ανθρώπων. Και με αυτό σε 400 περιπτώσεις. Οι συμμορίες είναι πολύ εθνοτικές, έχουν ιεραρχία, έχουν καλό δίκτυο, επιχειρηματικό χαρακτήρα, ψάχνουν την επόμενη ευκαιρία και παράσχουν πολλαπλού είδους υπηρεσίες με το χάρη ε, βρίσκουν ξενοδοχεία. Ε, ε, έχουμε λοιπόν κάποιους ειδικού αυτές οι συμμορίες των διακινητών ουσιαστικά εργάζονται στην παραοικονομία και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο έξυπνη, όχι μόνο γιατί πρέπει να καταστήλουμε αυτή την πρακτική, αλλά και σε έναν βαθμό πρέπει ουσιαστικά να ανταγωνιστούμε με αυτές τις τιμωρίες. Πρέπει να μειώσουμε τη ζήτηση και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να είναι ασφαλείς. Αν ε, κάποιος φτάσει στην Ελλάδα και φτάσει σε ένα hot spot, θα πρέπει να τον πείσουμε ότι ε, ουσιαστικά θα πρέπει να επαναχωρήσει από το συμβόλο που έχει με το διακίνητη, ο οποίος του έχει τάξει ότι θα τον βοηθήσει να φτάσει στη Γερμανία. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε την φυσική έλλειψη εμπιστοσύνη στα κράτη και στις κυβερνήσεις και ταυτόχρονα να τραβήξουμε τους ανθρώπους από δίκτυα που σχετίζονται με το πληθυσμό της διασποράς. Ουσιαστικά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ αποτελεσματικό δίκτυο διακινητών. Μπορούν να ε, σε πάνε από τέσσερι, σε τέσσερις μέρες από την Τουρκία στη Γερμανία. Το υπόσχονται και το πράττουν. Αυτή τη στιγμή δεν τους ανταγωνιζόμαστε. Ανέφερα τρία προβλήματα. Καταρχήν, πολύ λίγα κρατημέλη συμμετέχουν στη μεταγκατάσταση, στο μηχανισμό μεταγκατάσταση των προσφύγων. Αν ένα κράτος μέλος το οποίο θέλεις να φτάσεις ως μετανάστης, ως πρόσφυγας δεν συμμετέχει στο μηχανισμό με την κατάσταση δεν έχει νόημα καν να μπει στη διαδικασία. Δεύτερο, είμαστε υπερβολικά αργοί από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία, εργάζονται σκληρά να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν κάποιες αρχικές πρακτικές για το πώς θα ταυτοποιήσουν τους πρόσφυγες και ποιος πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το την κατάσταση. Ε, δεν είναι πολύ γρήγοροι ρυθμοί. Αντιμετωπίζουμε ε, πρακτικά προβλήματα, οι εμπορικές, αεροπορικές εταιρείες κάποια τη φορά θέλουν μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων να μεταφέρουν. Έτσι λοιπόν χρειάζεται περισσότερος χρόνος και το τίτλο το πρόβλημα νομίζω ότι είμαστε πολύ επιλεκτικοί στο τι κάνουμε. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε ανεθνικότητα, ή μόνοι που είναι επιλέξιμοι για τη μετακατάσταση πρέπει να έχουν 75% ποσοστό επιτυχία δηλαδή Σύριοι, Αφγανοί, Ιρακινοί, ενώ όλοι οι υπόλοιποι απορρίπτονται, αλλάζουν οι κανόνες ανάλογα με, τα γλωσσικά, με τις γλωσσικές δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο όπως είπα λοιπόν είναι πιο έξυπνο από εμάς και δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Δεύτερον, ποιες είναι οι κοινωνικές συνέπειες για τα Δυτικά Βαλκάνια εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Πρώτα απ' όλα είναι ένας αυξανόμενος φόβος μεταξύ των πληθυσμών ότι ε, θα εγκλωβιστούν εκεί, φοβούνται ε, τα, ε, τους συνοριακούς ελέγχους, ανησυχούν ε, για τα περιορισμένα ε, μονοπάτια μετακίνησης όπως για παράδειγμα το να έχουν ένα διαβατήριο φοβούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταματήσει να επενδύει ε, σε συνδέσεις μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια και δεύτερον βλέπουμε εντάσεις ανάμεσα σε αυτούς τους εγκλωβισμένους πληθυσμούς αλλά ε, και σε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, τα Δυτικά Βαλκάνια ως χώρες μετάβασης. Ε, πρόκειται για χώρες που έχουν σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, καθώς επίσης και μειονότητες που δυσχεραίνουν τα προβλήματα. Τρίτον, βλέπουμε αυξανόμενη πίεση για μετανάστευση από τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επικεντρωθεί στι ε, αιτήσει ασύλου που έχουν προτεραιότητα από τη Συρία. Βλέπουμε ε, ότι κάποιες χώρες έχουν να χειριστούν και αιτήσει από τα Δυτικά Βαλκάνια με αποτέλεσμα ε, η διαδρομή ασύλου να γίνεται πιο αλκιστική και με αποτέλεσμα να κάνουν και αυτοί αιτήσεις ασύλου αυτή η μετανάστευση είναι πολύ οργανωμένη, ε, διακόπτουμε τα μονομάτια εμβασμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε μια απώλεια πληθυσμού στις διάφορες ε, κοινότητες, πολιτικές κοινότητες των Δυτικών Βαλκανίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η, ε, η πολιτική εξουσία μειώνεται στις συγκεκριμένες περιοχές. Τρίτον, και θα τελειώσω με αυτό και συγγνώμη αν ε, ξέφυγα από το χρόνο μου. Τρίτον, όσον αφορά το, ε, τις πολιτικές συνέπειες, ε, πώς επηρεάζει η κατάσταση αυτή εκεί. Θα αναφέρω τρεις ιδέες. Πρώτον, συγκεκριμένα οι ε, σχέσεις στα Δυτικά Βαλκάνια γίνονται πιο δύσκολες. Η Σερβία είναι κεντρική όσον αφορά οποιαδήποτε διαδρομή διακίνησης ε, προσφύγων, όμως μικρότερες χώρες στην περιοχή. Δεν ξέρουμε πότε θα αλλάξουν και προς τα πού οι διάφορες πορείες με αποτέλεσμα να έχουμε μια βεβαιότητα. Η ε, Σερβία οπότε παίζει ένα βασικό ρόλο και πάντοτε υπάρχει ο... Ε, υπάρχει πειρασμός ε, όταν αναζητούνται νέοι, νέες διαδρομές. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και ιδιαίτερο όσον αφορά τι ε, σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα Δυτικά Βαλκάνια αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων ε, και τη συνεργασία που γίνεται όλο και πιο πολιτικοποιημένο και αυτή είναι η κατάσταση ιδιαίτερο στο Κόσοβο όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ε, πίεση διότι δεν έχουν σχέσει ελεύθερων θεωρήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι σιγά σιγά ο πληθυσμό αρχίζει να χάνει την εμπιστοσύνη ότι ποτέ θα αποκτήσει κάτι τέτοιο και αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα με τα σύνορα με το Μαυροβούνιο. Ε, η κατάσταση γίνεται πάρα πολύ πολιτικοποιημένη. Οι σχέσεις μεταξύ Κωσόβου και ε, της ε, Σερβίας ε, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αντιστρέφονται και σίγουρα η απελευθέρωση θεωρήσεων γίνεται όλο και πιο επιτακτική και τρίτον βλέπουμε ε, τα, την πολιτική σχετικά με την αναγνώριση ε, ετούντων ασύλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε κράτη-μέλη τα οποία είναι πιο σκεπτικιστικά σχετικά με την διεύρυνση ε, στην, ε, στα Δυτικά Βαλκάνια και είναι πιο, πιο διατεθειμένε αυτέ οι χώρε να παράσχουν άσυλο σε πρόσφυγε από τι συγκεκριμένε χώρε και από την άλλη χώρε οι οποίε υποστηρίζουν την διεύρυνση θέλουν να περιλάβουν τις χώρε των Δυτικών Βαλκανίων στι ασφαλεί χώρε Κλείνοντα με μια ιδέα θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει μπροστά της μια επιλογή μεταξύ αυτής της ε, λειτουργικής διάβρωσης ε, που δημιουργούν τα, οι διακινητές και οδηγεί σε μια κατακαιρμάτιση ή να αγκαλιάσει μια δυσλειτουργική ολοκλήρωση με τα Δυτικά Βαλκάνια και να συνεργαστεί πιο στενά με αυτές τις χώρες και βλέπουμε σιγά σιγά σημάδια προόδου όσον αφορά την προσέγγιση τους ε, στα δυτικά πρότυπα υποδοχής ε, και η ιδέα που έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη ιδέα να δημιουργηθεί κάτι παρόμοιο σαν το Δουβλίνο θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε αυτή την ενσωμάτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. και Καν. Ευχαριστώ καθηγητά. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, τι μπορεί να γίνει περαιτέρω για να βοηθήσουμε να σταματήσουν αυτές οι ροές. Άνθρωποι συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των προσφύγων με αποτέλεσμα ε, να έχουν τεράστια οικονομικά κέρδη από τον πόνο ανθρώπων ε, πώς θα βοηθήσει λοιπόν το να έχουμε μία μόνιμη οδό από αυτές τις παράνομες ώστε να περιορίσουμε τη ροή και ε, τέλος όσον αφορά την ε, αστάθεια που επικρατεί σε κάποιες χώρες πόσο ενέργεια πρέπει να ξοδέψουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε από αυτές τις αιτίε που επιφέρουν την αστάθεια και κάτι ακόμα που θα ήθελα να ακούσω είναι ότι γίνονται, πάρα ε, πολλές, γίνονται συζητήσεις σχετικά με αυτές τις ε, ροές προσφύγων και το κίνδυνο για την ασφάλεια. Πόσες αποδείξεις λοιπόν υπάρχουν για αυτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, αναφέρατε τη Ρουμανία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο εύξενος πόντος ίσως να μετατραπεί σε μία οδό μέσα από την οποία ε, θα μπορούν οι πρόσφυγες να καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε πολλά σχετικά με την περιοχή και για παράδειγμα πέρυσι ο αριθμός ε, των ε, προσφύγων από το Μαρόκο στην Ισπανία ήταν ε, το μισό σε σχέση με φέτος. Σήμερα υπάρχουν διπλάσεις στον εύξενο πόντο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι διακινητές θα μπορούν να μετακινηθούν εκεί και να ανοίξουν νέες διαδρομές μέσω της Ρουμανίας ή της Ουκρανίας ίσως. Και το δεύτερο θέμα είναι αυτή η παράνομη επιχείρηση, αυτή η οικονομία είναι ε, διεθνής, είναι διασυνοριακή και όταν βλέπουν λοιπόν ότι οι δυνατότητες είναι περιορισμένες σε μια χώρα, μετακινούνται αλλού. Αν λοιπόν είναι ενεργοί σε μια ακτή, πηγαίνουν κάπου αλλού για παράδειγμα δεν μπορούν, αν δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα σημείο τότε αλλάζουν ίσως το επιχειρηματικό τους μοντέλο αυτές οι τεράστιες συμμορίες που μετακινούνται μεταξύ χωρών. Σας ευχαριστώ. Πράγματι, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση άνευ προηγουμένου πρέπει να κάνουμε τα πάντα ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή να έχουμε αποτελεσματικά εξωτερικά σύνορα, να έχουμε τρόπους να διανέμουμε ανθρώπους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η πραγματική πρόκληση και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μου εγείρει ερωτήματα. Η πραγματική πρόκληση λοιπόν είναι να αξιολογήσουμε τι μέλη γενέστε. Ναι, φυσικά μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία με την Τουρκία ε, και ναι, σε αντάλλαγμα θα πάρουν χρήματα και ε, απελευθέρωση θεωρήσεων σε ως ανταλλάγματα. Μπορούμε να μαζέψουμε όμως κόσμο σε ένα τραπέζι στη Βιέννη για να επιλύσουμε το ε, πρόβλημα της Συρίας, για να σταματήσει η σύραξη εκεί. Ε, και να υπάρχει δυνατότητα για τους ανθρώπους να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Άμα όμως το κοιτάξουμε, 90 εκατομμύρια Αιγύπτιοι, 45 εκατομμύρια εξ αυτών επιβιώ, αγωνίζονται να επιβιώσουν καθημερινά. Αν λοιπόν έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα καράβι, τι θα κάνουν στη συνέχεια. Ε, στα ανατολικά, αν ο Πούτιν τρελαθεί και ε, προχωρήσει ακόμα πιο πολύ μέσα στην Ουκρανία και έχουμε άλλα 2 εκατομμύρια εκτοπισμένους, πού θα πάνε αυτοί. Οπότε είναι ερωτήματα αλληλεγγύης ε, τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε και θα πρέπει να τα θέσουμε με διαφορετικό τρόπο οπότε θα πρέπει ε, να έχουμε κοινέ προξεγγίσεις ε, και εδώ κριτικάρω και την ίδια μου τη χώρα. Μόλις πριν ένα χρόνο η Γερμανία δεν υποστήριζε μια, μια υποχρεωτική αναδιανομή διότι ήμασταν τόσο μακριά από όλο αυτό. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες πάντοτε αλλάζουν. Το ένα θέμα είναι λοιπόν να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους και οι παράλληλες ε, μερικές λύσεις ε, να ξεπεράσουμε την ε, σοβαρή πίεση. Νομίζετε λοιπόν ότι αυτό ευαρκεί είναι ένα ερώτημα πολιτικής βούλησης ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε και απίστευτα πράγματα όπως ε, για παράδειγμα να θέσουμε τον στρατό ανάμεσα στην Τουρκία και τα ελληνικά σύνορα και να απειλήσουμε ίσως ότι και θα γίνει βίαιος. Αυτό είναι κάτι που εγώ και κανένας από εμάς δεν επιθυμεί. Σας ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Σας ευχαριστώ με όλο τον σεβασμό στον Μάικλ Γκάλλος και το Ηνωμένο Βασίλειο το ένα θέμα αφορά τις ε, διμερείς ε, συμφωνίες ε, και την λεπτομερή εξέταση των προσφύγων που δεν πιστεύει επίσης σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ποσοστώσεων Όλο αυτό το σχέδιο λοιπόν είναι απαράδεκτο, έχει εφαρμοστεί από την, επιβληθεί από, την τη Γερμανία και από την καγκελάριο Μέρκελ να εφαρμόσει μια ε, πολιτική ανοιχτών θυρών και νομίζω ότι αυτό ήταν μια πραγματική καταστροφή όσον αφορά το ΣΕΝΚΕΝ. Τα δικά μου ερωτήματα είναι διάφορα. Πρόσφατα μου επιβεβαίωσαν ε, σε μια συζήτηση με τον ε, Μακεδόνο Υπουργό Εξωτερικών ότι ένας μικρός αριθμός ε, τζιχαντιστών που καταζητούνται έχουν ε, εισρεύσει σε αυτό το ε, ρεύμα προσφύγων και έχουν φτάσει στα Βαλκάνια μέχρι, όμως, να ταυτοποιηθούν όμως είχαν φύγει από τη χώρα και είχαν πάει στη Γερμανία, στη Σουηδία ή κάπου αλλού ποιος ξέρει. Το δικό μου ερώτημα είναι λοιπόν γιατί ε, δεν έχει ε, δοθεί πρόσβαση στην Europol, Eurojust και ούτω καθεξής ε, και γιατί δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα στις 24 ώρες με συνεργασία μέσω ενός υπολογιστή αντί να υπάρχει μια καταγραφή. Η ανταλλαγή λοιπόν πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ε, Δυτικής Ευρώπης ε, και το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωση, είναι, ε, είναι κάτι το οποίο δεν τα πάμε καλά σε αυτόν τον τομέα. Και πιστεύετε λοιπόν ότι το σύστημα Σέγγεν μπορεί να συγκρατηθεί όταν έχουμε αδύναμα εξωτερικά σύνορα, έχουμε πολιτικές ανοιχτών θυρών για τους πρόσφυγες, αλλά και κακές πληροφορίες ε, και υπηρεσίες αστυνόμευσης στον τομέα της ανταλλογής ε, πληροφοριών. Ε, άκουσα ότι υπήρχε ένας άντρας από το Μαδοβούνιο τον οποίο το στομάτησαν στα σύνορα στη Γερμανία και δεν ενημερώθηκε ποτέ η Γαλλία η Γαλλία ήταν ο προορισμός του. Και νομίζετε ότι η συνεδρίαση 51 της Γενέβης μπορεί να ισχύσει βλέπουμε ότι υπάρχουν ασφαλείς χώρες αλλά ε, αυτές, αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν τις πλούσιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης ε, διότι η συγκεκριμένη συνθήκη δεν είχε, εφαρμοστεί, δεν είχε σχεδιαστεί για τον σύγχρονο κόσμο και για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ θέλω να ρωτήσω καταρχάς, ε, το κύριο δίκτυο των μετακινητών τι εθνικότητα είναι, από ποια χώρα, δηλαδή σε ποια χώρα εδρεύει το πιο σημαντικό κομμάτι των διακινητών. Και το δεύτερο είναι ότι το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα παρατηρείται το εξή φαινόμενο. Ε, από τα νησιά περνάνε όλο και λιγότεροι πρόσφυγες που μιλούν Συριακά. Συγχρόνως, στα βόρεια σύνορά μας, στα Σκόπια, δεν επιτρέπεται να περάσουν πια παρά μόνο Σύριοι Αφγανοί και Ιρακινοί. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μείνει σε ένα σημείο που λέγεται σε μια περιοχή ειδωμένη και τώρα σιγά σιγά τους πάνε προς την Αθήνα. Αυτοί το επόμενο διάστημα θα πολλαπλασιάζονται. Τι μπορεί να γίνει με αυτόν τον κόσμο, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, διότι άλλο να μιλάμε για μερικές χιλιάδες και άλλο να μιλάμε σε λίγο καιρό για εκατοντάδες χιλιάδες. Thank you. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Συγγνώμη, ο κύριος Φρόιντ ήθελε το λέω. Περίμενε να μου ζητήσετε, να μιλήσω. Αυτή τη φορά δεν σήκωσα το χέρι μου και δεν μου ζητήσατε. Λοιπόν, έχω ένα δυο ερωτήσεις ε, οι οποίες αφορούν τον κατάλογο πραγμάτων στα οποία αναφερθήκατε κύριε καθηγητά και σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις εξηγήσεις. Οι επιχειρήσει διακίνηση οδηγούν σε πολιτικό και κοινωνικό κατακαιρματισμό στην περιοχή, είπατε περίπου στην αρχή. Αυτό ο πολιτικό και κοινωνικό ε, κατακαιρματισμό είναι εντό των χωρών, έτσι δεν αναφέρεστε στου πρόσφυγε. Αυτό το οποίο δεν ε, μπορώ να καταλάβω είναι ότι τονίζετε τόσο πολύ την ίδια την επιχείρηση διακίνησης που με οδηγεί στο ερώτημα δεν θα έρχονταν οι πρόσφυγες αν δεν είχε διακινητές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα συνέβαινε. Γνωρίζω ότι χρειάζονται τα σκάφη από την Τουρκία για να μπορέσουν να φτάσουν στα λυσιά, αλλά μέσα στην Ήπειρο, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, όπως έκανε και πολλοί, μπορούν να περπατήσουν έχουν και άλλους τρόπους ε, μεταφοράς και να, δεν χρειάζεται να εξαρτώνται τόσο πολύ από τους διακινητές. Τώρα, οι κοινωνικές συνέπειες ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Και πάλι, οφείλεται αυτό όλο αυτό το μεγάλο αριθμό προσφυγών. Οι περισσότεροι από αυτού δεν μένουν εκεί. Ελάχιστοι στην πραγματικότητα μένουν. Επομένω, τι κοινωνικέ ε, συνέπειε είναι αυτέ τι οποίε αναφέρεστε. Και τέλο, ή σχεδόν τέλος. Μήπως μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάτι το οποίο ακούσαμε σήμερα το πρωί από τον ε, υπονάβαρχο ο οποίος μας είπε ότι το 61% όλων των προσφύγων που διασχίζουν τα σύνορα από την Τουρκία στην Ευρώπη είναι Σύριοι. 61% και οι υπόλοιποι είναι Αυγανοί, Ιρακινοί και ούτω καθεξής. γεγονός το οποίο με εξέπληξε, διότι όταν εγώ μίλησα στον Υπουργό Εξωτερικών ε, ε, της Αυστρίας προσφάτως, μου είπε ότι μόνο ένα 20% των προσφύγων που περνούν από την Αυστρία είναι Σύριοι και ε, όταν το έψαξα είδα ότι δεν είναι 20% είναι 30% αλλά 30% είναι πάλι το μισό του 60%. Πού είναι, τι πάθανε οι υπόλοιποι στο μεταξύ. Και ε, τέλος θα ήθελα να πω και το εξής ε, προς τον κύριο Τάνοκ. Θεωρώ ότι είναι επονίδιστο και είναι πολιτικό παιχνίδι να εξισώνεται την περηφάνεια των μεταναστών με τις τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Παρίσι. Εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει καμία σχέση το γεγονός αυτό με τους πρόσφυγες. Πρόκειται για ανθρώπους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Παρίσι ή στο Βέλγιο. Ο κύριος Στάνοξ σχολιάζει εκτός μικροφών. Αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν Σύριοι ή αν ήρθαν από το Παρίσι, πήγαν στην ε, Συρία για να εκπαιδευτούν και επέστρεψαν στο Παρίσι. Δεν επρόκειτο για πρόσφυγες, μπορεί να χρησιμοποίησαν ε, ένα διαβατήριο, αλλά ακόμα και αυτό δεν είναι βέβαιο, γιατί εγώ δεν εμπιστεύομαι όσα διαβάζω πουθενά πλέον. Ευχαριστώ. Οι τελευταίες σας παρατηρήσεις ε, ε, πραγματικά νομίζω ότι έρχονται να ε, μας εκπλήξουν διότι είστε δημοσιογράφος. Ε, είναι αργά το απόγευμα και πραγματικά αυτό που μας λέτε είναι φρικτό για την έντυπη δημοσιογραφία. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε δύο θέματα και να θέσω και εγώ μια ερώτηση. Πρώτον, πρώτη φορά στη διάρκεια της αποστολής μας ε, στα τέλη Σεπτεμβρίου στο Northwood όπου είχαμε μεταβεί για να δούμε τις ε, διαδικασίες της επιχείρησης Αταλάντη Εκεί λοιπόν μας εξήγησαν τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα των πειρατών. Και επειδή είμαι οικονομολόγος, με άγγιξε ο τρόπος αυτός με τον οποίο μας τα εξήγησαν. Και κάποια άλλα μέλη επίσης, κάποια άλλοι ευρωβουλευτές και αυτοί ευαισθητοποιήθηκαν ως προς τα όσα μας είπαν. Ε, Ε, και μάλιστα κάποια στιγμή μα είπαν ότι ε, πήγαν λίγο παραπέρα και μα είπαν ότι εμεί έχουμε να ανταγωνιστούμε αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα. Και ο μόνο τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι να αντιδράσουμε και να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα. Ε, είμαστε βέβαια λίγο πιο μεγάλοι, ελπίζω, πιο σημαντικοί παράγοντες Μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα για τις ε, πιθανές απειλές ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας συγκλονίζουν όλους, αλλά πρέπει να τα αξιολογήσουμε εμείς όλα αυτά. Εμείς είμαστε υπό Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσον υπάρχει ακόμα και δυνητικός ε, σύνδεσμος Ακόμα και ο ελάχιστος πιθανός σύνδεσμος είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξερευνήσουμε διότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τις πιο ζωφερές εκδοχέ. Δεν μπορούμε απλώς ε, να παραβλέψουμε κάποια πράγματα γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια απειλή. Ε, θεωρώ ότι αποτελεί λανθασμένη νοοτροπία αυτό, επομένως θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε μια αξιολόγηση και να αξιολογήσουμε και αυτά τα ενδεχόμενα. Και ακόμα και αν λέτε ότι κάποιοι γεννήθηκαν στο Παρίσι και μετά ε, πήγαν να εκπαιδευτούν στη Συρία, στο Ιράκ ή κάπου αλλού, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κατά πόσον ε, μπορεί να ήταν και Γάλλοι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ήταν κάποιος ε, ε, υπήκος, το συνέβη και στην Πολωνία, το είδαμε και στο Λονδίνο. Ε, στις, ε, στα γεγονότα πριν από 10 χρόνια περίπου, 8 χρόνια πιο συγκεκριμένα, με ανθρώπους που είναι άνθρωποι δεύτερης γενιάς ε, και έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί. Ε, πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τα θέματα αυτά και την εσωτερική ασφάλεια. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μου παρατήρηση και η δεύτερη παρατήρησή μου είναι για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρέπει να ξεχάσουμε δηλαδή τη διαδικασία της Θεσσαλονίκης λόγω αυτής της λειτουργικής διάλυσης. Μήπως θα έπρεπε να τα ξανασκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο ώστε να μην επέλθει από σύνθεση. Για παράδειγμα, ε, όταν εξετάζουμε το άσυλο ε, θεωρούμε δεδομένο ότι πρόκειται για αποτυχημένα κράτη ε, που δεν ισχύει πάντα για όλες τις περιπτώσεις δεν είμαστε ε, ακόμα σε θέση να το πούμε για τα περισσότερα κρατημέλη. Και φυσικά ε, κάποιες χώρες πιέζονται πολύ περισσότερο λόγω ε, του γεγονότος ότι οι περισσότερες μεταναστευτικές ροές περνούν από τα Δυτικά Βαλκάνια. Αλλά και στη διάρκεια του πολέμου ο αριθμός των ανθρώπων που ήταν διατεθειμένοι να μεταναστεύσουν δεν ήταν τόσο υψηλός όπως μας είπατε κι εσείς. Επομένως, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για την αλλαγή αυτή. Ε, ήταν ε, ίσως το γεγονός ότι φαντάζονταν ότι θα τους απελάσουν ή ότι δεν θα, θα τους αποκλείσουν από τη διαδικασία της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ε, Ο κύριος Κάμπελ Μπάνεμαν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα προς ενημέρωση προς τον κύριο Φρόιντ εδώ μπροστά. Να σας πω ότι είχα ε, ενημέρωση από τους πεσμεργά για θέματα ασφαλείας και για τους Ισραηλινούς συμμετέχω στη σχετική αντιπροσωπεία και, και οι δύο μα λένε ότι υπάρχουν παριστρήσει αυτών των προσφύγων που φτάνουν στην Ευρώπη. Και εγώ δεν διαβάζω εφημερίδε, ε, είναι από μυστικέ υπηρεσίε οι πληροφορίε που έχω και πραγματικά είναι πολύ ε, σοβαρή απειλή, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορείτε να το αρνείστε. Χρησιμοποιήθηκε ένα διαβατήριο από 8 διαφορετικού ανθρώπου και ένα εξ αυτών ήταν τρομοκράτη. Δεν μπορούμε να είμαστε ε, έτσι αδρανεί και να τα ε, ε να απαξιούμε για όλα αυτά που ακούμε. Ξεκινά ένα διάλογο μεταξύ δύο συναδέλφων. Κύριε Γκάλερ, άμα θέλετε να απαντήσετε, μπορείτε να ζητήσετε το λόγο. Όχι. Καλά. Ο κύριο Καν. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί γίνεται. Η διαφορά όμως και το επιχείρημα το οποίο προσπαθούσε να αναπτύξει ο συνάδελφος είναι ότι υπάρχουν πρόσφυγες τους οποίους πρέπει να δείξουμε κατανόηση και μετά υπάρχουν και εγκληματίες οι οποίοι παρισφρίουν στα διάφορα ε, προσφυγικά ρεύματα και υπάρχουν πάντα διάφορες διαδρομές είτε υπάρχουν πρόσφυγες είτε όχι. Ανέκαθεν το έκαναν. Επομένως εμείς ως κοινωνία πρέπει να έχουμε προηγμένα συστήματα που θα μπορούν να αντιληφθούν και τα δύο και επομένω πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του εγκληματίε. Και αυτή είναι η ουσία. Ο κύριος Έλλης. Θα προσπαθήσω να επανέλθω στο ζήτημα. Υπάρχει αυτός ο φόβος ότι θα συνδεθεί η μετανάστευση με την τρομοκρατία. Όπω είπατε σωστά, υπάρχουν κάποιες πηγές από το Ισραήλ και πηγές που ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνο όμως από ένα σκοπό μόντου οπεράντη δεν θα ήταν ε, εντελώ ε, εξωτικό να ξεκινήσει κάποιος ε, στη Μέση Ανατολή να διαστήσει την Τουρκία, τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και να φτάσει στον τόπο που θέλει να δράσει. Δηλαδή, με πρακτικούς όρους, αν θε να είσαι αποτελεσματικό ω τρομοκρατική οργάνωση, μπορείς να διαλέξεις πολύ εύκολα άλλου τρόπους να βάλεις ανθρώπους στην Ευρώπη ή να ενεργοποιήσει ανθρώπους εντό τη Ευρώπη, Για να προβούν σε οποιαδήποτε είδου επίθεση. Προφανώς υπάρχουν διάφορες πηγές που ψιθυρίζουν για το θέμα αυτό. Όμως ε, δεν ε, είναι απαραίτητο ε, να χρησιμοποιηθούν οι πρόσφυγες ως πρόσφυγες να μπουν στην Ευρώπη για να επιτεθούν. Δηλαδή ουσιαστικά πέρα από τον κύριο κίνδυνο ότι οποιοδήποτε έρθει στην Ευρώπη μπορεί ως ένα βαθμό να έχει κάποιες ε, τρομοκρατικές ε, προθέσεις. Ε, πρέπει να αξιολογήσουμε και το τι λένε αυτές οι πηγές. Πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνω ολοκληρώνεται η διαδικασία των ρωταπαντήσεων απαντήσεων και θα ήθελα να απαντήσει ο κύριος Πάρξ στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τις εξαιρετικές ερωτήσεις. Είναι πολλές. Ε, τις ομαδοποίησα σε τρεις προσεγγίσεις. Καταρχήν νομίζω ότι θα λέτε μεγαλύτερη ακρίβεια για τη φύση του προβλήματος. Θα αναφερθώ πρώτα σε αυτό. Κατόπιν τη φύση της εσωτερικής μας απάντησης και την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες. Για τη φύση του προβλήματος καταρχήν. Θα ξεκινήσω με την οδό από τον Αυξήνο Πόντο, γιατί είναι το πιο εύκολο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ κερδοφόρο. Υπάρχουν εκθέσει ότι έχουμε ένα-δύο σκάφη που ακολουθούν αυτή την οδό. Ακόμη βέβαια δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, αλλά δεν έχουμε στραφεί, στρέψει εντατικά τι έρευνε μα προ αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν άλλε οδοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη μετανάστευση. Βέβαια, τώρα αυτό μα οδηγεί στην ερώτηση πόσο διεθνικά είναι αυτά τα δίκτυα των διακινητών. Τίνουν να βασίζονται σε υφιστάμενα ε, εγκληματικά διασυνοριακά δίκτυα. Έτσι, λοιπόν, ε, ξέρετε ότι υπάρχει η οδός της Ουκαΐνης, είναι σταθερή αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η οδός του λαθρεμπορίου όπλων. Όμως, ε, καταρχήν θα αποφύγουν τη συνεργασία με τους ε, ίδιους παίκτες, ε, κυρίως με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, όμως σε δεύτερο επίπεδο πάρα πολλά συμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, αν μια χώρα κλείσει τα σύνορά της και πρέπει οι μετανάστες να περάσουν βουνά και δάση, τότε απλώς οι ντόπιοι θα δράξουν αυτή την ευκαιρία. Αυτό σε σχέση λοιπόν με το διασυνοριακό χαρακτήρα. Τώρα για τους συνδέσμους με την τρομοκρατία. Είμαι πολύ προσεκτικός απέναντι στο θέμα αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε ως συγκεκριμένη απειλή είναι ότι μπορούμε να δούμε Ευρωπαίους ξένους μαχητές να ξαναέρχονται και να ξαναμπαίνουν στην Ευρώπη με προσφυγικές ροές. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν νόμιμο τρόπο να ξαναμπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τους παρακολουθούμε και μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται, να έχουν παρισφρήσει σε αυτές τις ροές. Και δεύτερον υπάρχει και ένα σύνδεσμος με τον πληθυσμό της διασποράς. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλες ε, κοινότητες ε, και εκεί η εισρωή δημιουργεί εντάσεις αλλά από όσα μαθαίνω δεν είναι σαφή τα πράγματα δεν έχουμε σαφή εικόνα για παραδείγματο χάρη τι θέλει να πετύχει το Ισλαμικό κράτος. Δηλαδή στο αν προσπαθεί ακριβώς να καταφερθεί κατά της φιλοξενίας μας ή της μεταναστευτικής στρατηγικής μας. Εγώ νομίζω ότι λογικά θα ενεργοποιήσει ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ. Εγώ δεν έχω το επίπεδο της δικής σας πληροφόρησης. Τώρα, για τον αριθμό των σύρων. Πολύ ψηλοί μου ακούγονται αυτοί οι αριθμοί. Πρέπει να έχουμε κατά νου το πόσο πολύπλοκος είναι ο κόσμος γύρω μας. Και αν το έχουμε αυτό κατά νου, μιλάμε για σχετικά μικρή αναλογία. Πολύ μικρότερη από ό,τι θα πίστευε κάποιος. πρόσφατα το ότι έχουμε Σύρους, Ιρακινούς και Αφγανούς ε, και Όλοι αυτοί αποτελούν το 1 τρίτο των αιτήσεων ασύλου που κατατίθεται. Νομίζω τώρα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα έχουμε φτάσει στα 2 τρίτα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Νιγηριανή νομίζω είναι η εθνικότητα. Στην Ιταλία άνθρωποι από την υποσαχαρή Αφρική. Στην Πολωνία Ουκρανοί. Έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση λοιπόν. Αυτό σε σχέση με το ποιο έρχεται και τη φύση του προβλήματος. Τώρα, για τη φύση της εσωτερικής απάντησης και τη συνεργασία με τους κοντινούς μας γείτονες. Υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις για μία απάντηση από τις διοκτικές αρχές, συνεργασία με τις διοκτικές αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Κατά ένα νόημα, εδώ έχουμε ουσιαστικά ένα πρόβλημα πολύ συχνά η Τουρκία και άλλες χώρες ε, ε, ξέρουν ότι εμείς είμαστε κάπως διστακτικοί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για τρομοκράτες λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων και θέλουν να μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες για τους δεχτούμενους εταίρους, όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση Θεωρείται ότι είναι δύσκολο κάτι τέτοιο και για τα Δυτικά Βαλκάνια και οι διοκτικέ αρχές όταν θέλουν να λειτουργήσουν ω τέτοιε, είναι, έχουν πολύ ισχυρό ρόλο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την καταπολέμηση τη τρομοκρατίας αυτό το κάνουν πολύ αποτελεσματικά από όσο βλέπουμε. Όταν μιλάμε ε, τώρα για την διακίνηση, ε, για το λαθρεμπόριο, λιγότερο. Δηλαδή έχουμε κάποια σημεία επί το οποίο θεωρητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά είναι κάπω δύσκολο το ζήτημα. Τώρα για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσω αυτό είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει. Παραδείγματο χάρη, πολλά κράτη-μέλη έχουν αξιωματικού συνδέσμου μετανάστευση στην Τουρκία και σε άλλε χώρε. Όλοι προσπαθούν να οικοδομήσουν επαφέ και να έχουν μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Τώρα μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να του βοηθά να συνομιλήσουν μεταξύ του. Ήταν εξάρτητα δρούσαν. Τώρα η Frontex έστειλε ένα δικό τη αξιωματικό σύνδεσμο στην Τουρκία. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί νωρίτερα. Γιατί είχε την αρμοδιότητα. Έτσι λοιπόν σας αυτός ο τρόπο να κινηθούμε στο μέλλον. Δηλαδή να οικοδομήσουμε τις ικανότητές μας. Το θέμα των ε, νομικών οδών, αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε. Κοιτάξτε τώρα, πώς να ανταγωνιστούμε με τις ε, διακινητές. Εσεί ε, είπατε αυτά τα λόγια, λέει πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι, εγώ χρησιμοποίησα αυτά τα λόγια και θέλω να με κατανοήσετε εύκολα. Μερικέ φορέ πρέπει να πλουστεύει κανεί. Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε εκεί όπου μπορούμε. Όπω είπα στην εισαγωγή μου, πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά και να μπορούμε να οδηγούμε του ανθρώπου σε ασφαλεί συνθήκε όπου μπορούμε και να του δίνουμε κάποιε μακροπρόθεσμε οδού. Δεν ξέρω το αν δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χάρη να έχουμε απαλλαγή της υποχρεώσης θεώρησης για τους Ερυθρέους. Φαντάζομαι ότι και αυτό θα επιφέρει κάποιε δυσκολίε και καθυστερήσει, αλλά αν παρουσιάσουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, να πούμε αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, εκεί που ζείτε έχετε κάποια δυσευκαιρία, έτσι λοιπόν, ε, δυσευκαιρία, έτσι λοιπόν έχουμε ένα μείγμα ε, ανταγωνιστική απάντηση, αλλά και δημιουργίας νομικών οδών. Αυτό για την εσωτερική απάντηση. Και αν έχω χρόνο, πολύ γρήγορα, να αναφερθώ και στο τι μελιγενέστε. Υπάρχουν πολλέ εκκλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση για τη μετανάστευση. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι καθυστερημένο σύστημα μετά από φαινόμενο όπως η Αραβική Ένωση που περιμέναμε 400.000 άτομα και δεν ήρθαν και τώρα ήρθαν. Τι εξηγεί λοιπόν αυτό το χάσμα, αυτό το κενό μεταξύ της αρχικής, του αρχικού ξεσπάσματος της σύγκρουσης, της σύραξης και το πότε έρχονται οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά που παρεμβαίνουν. Μετά την Αραβική Ένωση πολλοί άνθρωποι επέστρεψαν στην περιοχή γιατί ήλπιζαν σε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έρχονταν εδώ. Υπάρχουν πολύπλοκοι παράγοντες. Θα το δείτε και με την Ερυθρέα αυτό. Αν πιέσουμε την Ερυθρέα ε, ουσιαστικά να αλλάξει τα πράγματα τότε, ε, εκεί ε, βλέπετε ότι έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό ανδρών που δεν αποτελεί έναν κινδύνο ασφαλείας. Δεν το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν όχι σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το αντίστροφο και για τη συνθήκη της Γενέβης. Ειλικρινά, σκέφτομαι πώς θα επικαιροποιήσουμε όλο το σύνολο των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μα Τα τελευταία 25 χρόνια λειτουργούσαμε βάσει μιας ιδέα ότι όλα συμπλέουν προς ε, φιλελευθερέ δημοκρατίες και εμεί στη Δύση μπορούμε να προσφέρουμε μια προσωρινή προστασία σε ανθρώπους που είναι σε κίνδυνο. Επειδή θα αυτοδροπηθούν οι χώρε αυτέ, θα επιστρέψουν. Είναι πάντα λοιπόν προσωρινή η κατάσταση και θα οικοδομήσουμε άλλε χώρε για να φιλοξενήσουν μετανάστε. Νομίζω ότι όμω τώρα είμαστε σε ένα παράδοξο ότι άλλε χώρε γίνονται πιο πλούσιε, με καλύτερα ε, με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης αλλά δεν γίνονται πιο φιλελεύθερες. Λοιπόν δεν είναι στην ίδια θέση με την οποία είμαστε εμείς για να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες και δεν φαίνεται οι άνθρωποι να θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα του, γιατί δεν πιστεύουν ότι θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να κατακαιρματίσουμε τις ε, ιδέες της Δυτικής Ευρώπης και να προωθήσουμε να, τα άλλα κράτη την ιδέα να δημιουργήσουν τα δικά τους συστήματα φιλοξενίας ανθρώπων. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλους τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας τους υφιστάμενους μηχανισμούς. Και δεν θα πρέπει να έχουμε ιερά ανέγγιχτα πράγματα. Σας ευχαριστώ. One remark. Επιτρέψτε μου ένα ε, σχόλιο προς τον κύριο Γκάλερ. Ξέρω, εδώ ε, και, εδώ και 1,5 χρόνο ε, είμαι ευρωβουλευτής. παλαιότερα ήμουν βουλευτής το ε, Πολωνικό Κοινοβούλιο και από τότε συμμετείχα στις επίσημες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου που αξιολογούσαν ε, το μεγάλο σχέδιο για ε, την ε, φιλοξενία των προσφύγων σε περίπτωση που γινόταν κάτι στην Ουκρανία. Ναι, υπάρχει ποικινομορφία, όμως ακόμα υπα, επαφίεται στα κράτη-μέλη ως να κάνουν αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ. Και εδώ λύγει αυτό το κομμάτι της, της ατζέντα, της ημερήσιας διάταξης. Σας παρακαλώ μην αποχωρήσετε διότι τώρα θα περάσουμε σε μια ακαδημαϊκή αξιολόγηση σχετικά με την ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 και ο μιλητής μας ε, είναι ο καθηγητής Αλεξάνδρου ε, Ματιλέρα από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Σας ευχαριστώ. Και πάλι κυρίες και κύριοι, ε, παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, καθηγητή Αλεξάνδρ Μάτλερ, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τις ε, νομικές συνέπειες της ενεργοποίησης της πιθανές συνέπειες της ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 της συνθήκης. Καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ ε, πολύ για την εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βεβαίως όταν παρουσιάζεται ένας ομιλητής με τα λόγια ακαδημαϊκή παρουσίαση σίγουρα νιώθουμε ένα αίσθημα στην αίσθηση στην αίθουσα ε, ανησυχίας, όμως δεν νομίζω ότι έχουμε έρθει εδώ για κάτι ακαδημαϊκό ε, και θεωρητικό. Ε, πρόκειται για πρακτικά ζητήματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί ύστερα από ε, μία σειρά τραγικών γεγονότων Βεβαίως είναι το αποτρόπαιο έγκλημα ε, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και έχει σοκάρει όλους μας και ακόμα νιώθουμε τις συνέπειες των όσων έχουν συμβεί και το νιώθουμε και εδώ στις Βρυξέλλες απευθυνόμενος ε, στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της ε, Γαλλίας χαρακτήρισε τα γεγονότα αυτά ως ε, εγκλήμα, ως ε, πράξη πολέμου και έδωσε την εντολή στον Υπουργό Αμήνης του ε, να πάει στις Βρυξέλλες και να ενεργοποιήσει το άρθρο 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα να τεθεί το ερώτημα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια βρισκόταν σε πόλεμο και αν ναι τότε πώς θα πράξει αυτό το πόλεμο και προς έκπληξή μου θα πρέπει ε, να ε, παραδεχτώ ότι ε, το Συμβούλιο Υπουργών Αμήνης και Εξωτερικών εξέφρασαν ομόφωνα την υποστήριξή τους στη Γαλλία και την ετοιμότητά τους να παράσχουν όλη την αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη και ναι αυτό, αυτά είναι τα λόγια από τα πρακτικά της συνεδρίασης. Θα πρότεινα ε, λοιπόν να ε, διαρθρώσω την ομιλία μου και την παρουσίασή μου σε τέσσερα μέρη. Πρώτον, ε, ένα γενικό κομμάτι σχετικά με τα μέτρα τα οποία μπορούν να λυμφθούν στα πλαίσια του άρθρου 42.7. Δεύτερον, θα ήθελα να μοιραστώ τις απόψεις μου σχετικά με τη διαδικαστική πορεία με την οποία τα κράτη-μέλη έχουν κινηθεί σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τρίτον, θα σας ε, ενημερώσω ε, σχετικά με το τι στρατιωτική υποστήριξη μπορούν να προσφέρουν οι εταίροι στη Γαλλία και τρίτον, και τέταρτον συγγνώμη, θα μιλήσουμε για μια ανταπόκριση που, που δεν αφορά μονάχα τα στρατιωτικά μέσα αλλά αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Συνοχή και αλληλεγγύη. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω σκεπτόμενοι λιγάκι το άρθρο 42,7. Υπήρξαν ε, διάφορα ε, σχόλια σχετικά με το ότι για ποιο λόγο η Γαλλία δεν ενεργοποίησε το άρθρο 5 της συνθήκης της Washington δεν νομίζω ότι αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη διότι από την εποχή του Σαρτεγκόλ η Γαλλία είχε μια δύσκολη σχέση με την ιδέα του να ε, εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εθνική της ασφάλεια. Όμως ε, το ενδιαφέρον κομμάτι αφορά το ότι άμα εξετάσουμε ε, το τα λόγια πώς είναι γραμμένα τα δύο άρθρα, το 42,7 αναφέρει συγκεκριμένα ότι είναι, είναι πιο αυστηρό, είναι πιο συγκεκριμένο διότι σε περίπτωση επίθεσης τότε τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να παράσχουν βοήθεια με κάθε μέσο ε, που έχουν στις δυνάμεις τους, ενώ από την άλλη ε, η συνθήκη της Washington λέει ότι θα πρέπει ε, ο εταίρος να βοηθηθεί με όποιον τρόπο θεωρείται ο καλύτερος. Βεβαίως ε, και τα δύο άρθρα ήταν διπλωματικές υποσχέσεις ε, και έτσι λοιπόν δεν σημαίνουν αυτά αυτά ε, κάτι το ιδιαίτερο. Η μόνη διαφορά με το άρθρο 5 είναι ότι η συνθήκη της Washington έχει ένα απτό πακέτο στρατιωτικών μέτρων ενεργές μονάδες ε, του ΝΑΤΟ, ακόμα ε, και δυνατότητα διαμοιρασμού των ε, πυρηνικών αποθεμάτων. Και όλες αυτές οι υποσχέσεις με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα της συμμαχίας να ανταποκριθεί σε μια επίθεση. Από την άλλη τώρα, το άρθρο 42.7 δεν έχει την ίδια αξιοπιστία, όμως δίνει κάτι σαν λευκή επιταγή. Αυτό που σημαίνει δηλαδή το ότι τα πάντα εξαρτώνται από ε, το τι θα προσφέρουν ε, σε αυτή την επιταγή τα κράτη-μέλη. Δηλαδή ε, ο καθένας μπορεί να πάρει και να προσφέρει ό,τι θέλει. Και αυτό είναι που θα απασχολήσει και το υπόλοιπο της παρουσίασής μου. Στην εισαγωγή μου ανέφερα ήδη ότι με εξέπληξε ο τρόπος ε, με τον οποίο ενεργοποιήθηκε το άρθρο ή δεν ενεργοποιήθηκε ανάλογα με το πώς, θα πρέπει να, πώς θέλετε να το ε, αντιληφθείτε. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση ήταν ε, κάπως ελαφρά παρμένη και αυτό αφορά αφενός το γεγονός ότι, μια προηγούμενη ότι δεν υπήρχε μια επίσημη απόφαση του ε, Συμβουλίου και ε, διότι λέγεται ότι καμία επίσημη ε, απόφαση του Συμβουλίου δεν απαιτείται για να ενεργοποιηθεί και αυτό φυσικά είναι γρήγορο και ευέλικτο, όμως ταυτόχρονα οδηγεί και σε ένα νομικό κενό πέρα από το γεγονός ότι το άρθρο αναφέρεται ε, στο άρθρο 51 του ΟΗΕ σχετικά με την αυτοάμυνα, όμως τώρα το να χρησιμοποιήσει την αυτοάμυνα ως αίτια πολέμου, πάρα πολλές ε, χώρες ε, μαζί και η Γαλλία έχουν βομβαρδίζουν εδώ και μήνες το ISIS, οπότε θα απαιτούνταν κάποια επιχειρηματολογία και η επιχειρηματολογία μπορεί να τεθεί, όμως δεν συνέβη ε, και έτσι είμαστε σε δύσκολο έδαφος από νομικής άποψης. Δεύτερον ε, και ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι συμφωνήθηκε σε, επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης και θα έλεγα ότι το άρθρο 42.7 αφορά την κοινή άμυνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πηγαίνει σε πόλεμο. Έτσι λοιπόν θα ήταν ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει το Συμβούλιο διότι η επικήρυξη ε, πολέμου είναι, αν δεν είναι αυτό κάτι που αφορά το Συμβούλιο τότε τι είναι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, όσον αφορά τη συζήτηση για το 42-7 σε επίπεδο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, σημαίνει παραδόξως ότι δεν μιλούμε πραγματικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση που πηγαίνει σε πόλεμο, αλλά στην πραγματικότητα για τους ευρωπαϊκούς εταίρους που προέρχουν βοήθεια στην Γαλλία για να κάνει το δικό της πόλεμο. Τρίτον, όπως υπογραμμίστηκε από την ύπατη εκπρόσωπο, η διαδικασία αυτή αφορά την ενεργοποίηση διμερούς ενεργασίας και βοήθειας και αυτή η προτίμηση για διμερείς λύσεις ε, είναι φυσικά κατανοητή εν ώψη των όσων ανέφερα προηγουμένως όμως ταυτόχρονα κατά τη γνώμη μου αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε στις θέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου πριν από 14 χρόνια με την στρατιωτική της δηλαδή ανταπόκριση. Η απάντηση λοιπόν ε, το, ε, της 11 Σεπτεμβρίου αποτελούσε ενότητα ε, σκοπού και αυτό ε, το έγινε το 2009-2010 δηλαδή 8-9 χρόνια αργότερα και τότε ο πόλεμος στο Αφγανιστάν ε, ήδη είχε πάρει ε, μια στροφή προς το χειρότερο και δεν ξέρω αν μπορούμε να αντέξουμε μια τέτοια αλλαγή άλλη μια φορά. Ε, τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα τι είδους βοήθεια μπορούν να παράσχουν οι ευρωπαϊκοί εταίροι προς την Γαλλία και εδώ θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στην στρατιωτική υποστήριξη και από την άλλη τη μη στρατιωτική υποστήριξη όσον αφορά την ε, μάχη κατά της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, κάτι το οποίο ξεπερνά τα όσα ε, καλύπτει το άρθρο 42.7 διότι αυτό εν τέλει αφορά ε, τα θέματα κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Όμως όσον αφορά τώρα τον στρατιωτικό παράγοντα Και φυσικά το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι η στρατιωτική υποστήριξη στην ε, Operation Μασάλ ε, και στην ε, διεθνή συνεργασία κατά του ΝΤΑΕΣ, του Ισλαμικού κράτους. Και φυσικά αυτό σημαίνει δυνάμεις για να εντετικοποιηθεί η στρατιωτική εκστρατεία, ιδιαίτερως όσον αφορά τις ε, δυνατότητες ε, για να υπάρξουν περισσότερες επιθέσεις. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ε, η εκστρατεία κατά του ISIS ήταν μία αποαέρος εκστρατεία που είχε να κάνει με την διαθεσιμότητα των στόχων. Το μπορεί να περιλαμβάνει όμως ε, και ε, ναυτικά εφόδια. Κάποιες ε, χώρες ήδη συνοδεύουν το Charles de Gaulle στην Μεσόγειο ή σκοπεύουν να το κάνουν μελλοντικά. Και σε περίπτωση που η περιοχή του Λεβάντα γίνει μια περιοχή που δεν θα είναι φιλόξενη εξαιτία της εισδοχής ε, ε, ανεπτυγμένων ε, συστημάτων αέρος, τότε η υποστήριξη μπορεί να αυξηθεί και να περιλαμβάνει κάθε είδους στρατιωτικό εξοπλισμό. Και η τρίτη διάσταση που αφορά το θέμα αφορά τη χρήση ειδικών δυνάμεων τόσο για, ε, στο, για επιθέσεις όσο και για στρατιωτική υποστήριξη ε, στις ε, τοπικές δυνάμεις και φυσικά οι συζητήσεις αυτές μεταξύ της Γαλλίας και των εταίρων έχουν ξεκινήσει σήμερα λάβαμε νέες ειδήσει σχετικά με την γερμανική προσφορά να αποστείλει και αυτή βοήθεια, μια φρεγάτα και όσον αφορά την εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους αφορά και ε, την βοήθεια ε, προς τη Γαλλία σε άλλα ζητήματα έχουμε τις ε, αποστολές Σαμάλ Μπακάν και Σοφτινέλ που θέτουν τεράστια πίεση στην ε, Γαλλία το Μπαχκάν έχει 3.000 πληθυσμό, η Σοκτινέλ 10.000 σε γαλλικό έδαφος και αυτές είναι μονάχα οι μεγάλες εκστρατείες, υπάρχουν και άλλες μικρότερες που προστίθενται σε όλο αυτό. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο ασκεί μεγάλη πίεση ε, στις γαλλικές δυνάμεις. Δεν τη φτάνουν στα όρια της ε, βέβαια, όμως ε, υπάρχει μεγάλη πίεση όσον αφορά τις γαλλικές δομές ε, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να το συντηρήσουν για πάρα πολύ καιρό ακόμα εκτός εκτός και αν ε, στρατολογηθεί νέο προσωπικό όμως ε, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να υποστηρίξουν την ε, Γαλλία υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ ε, που είναι διαθέσιμες όπως είναι για παράδειγμα μια εναλλακτική στο πλαίσιο του ΟΗΕ, στο Λίβανο, στο Μαλί. Και τώρα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι αυτό προσφέρει και μια ευκαιρία για να ξανασκεφτούμε την παρούσα, ε, την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην περιοχή του Σαχέλ που είναι αρκετά μεγάλη όμως κατατιμισμένη ε, όσον αφορά την θεσμική της οργάνωση Οπότε, αν θέλουμε μια ευρύτερη πρόταση για ποιο λόγο να μην ενισχύσουμε ε, την, ε, τις δραστηριότητες ε, της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εκστρατεία όπως για παράδειγμα η στρατηγική του Σαχέλ πριν από τέσσερα χρόνια. Επίσης θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας μέσω πληροφοριών, αστυνόμευσης και δικαστικής συνεργασίας, διότι όσον αφορά την ε, απειλές της τρομοκρατίας στις ευρωπαϊκές πόλεις, εκεί έγινε η πραγματική συζήτηση και κατά την άποψή μου πρόκειται επίσης και για έναν ε, τομέα ε, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία για τον εξής απλό λόγο. Κατ' εμέ, η εσωτερική αγορά δεν θα λειτουργήσει πραγματικά εάν δεν υπάρχει πραγματικά, ε, πραγματική αυθεντική εσωτερική ασφάλεια. Αυτό είναι η όλη ουσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κυρίως ε, εάν ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίσουν όλο και περισσότερο να θέλουν να παρισφρήσουν στη Σέγγεν για λόγους ασφαλείας. Ε, δεν είμαι βέβαια η Δήμων σε θέματα ιστορικής ασφαλείας, αλλά ε, με εκπλήσει το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει γενικότερα έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χώρο Σέγγεν και ε, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την ε, διαστραβρούμενη συλλογή πληροφοριών από τη Σέγγεν αστυνόμευση και δίωξη στη συγκεκριμένη περιοχή. Ε, και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει και η ίδια η Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, για την ενίσχυση των συνόρων αλλά και για όλες τις υπόλοιπες πτυχές ε, κυρίως. Θα χρειαστούμε σίγουρα κάποια περισσότερα εργαλεία διότι δεν πιστεύω ότι εάν βασιστούμε στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συστημάτων και μόνον θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια λύση. Υπάρχει επίσης και ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ακριβώς ε, διότι το άρθρο αναφέρεται σε όλα τα μέσα στη διάθεση των κρατών μελών και φυσικά η συζήτηση αυτή ε, θα πρέπει να αφορά τα πάντα, είναι αναπόφευκτο και φυσικά αυτό είναι κάτι που και ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος έκανε ε, συνδέοντας τις συνέπειες για τον προπολογισμό, για την απαιτούμενη απάντηση που πρέπει να δοθεί σε θέματα ασφαλείας με μακροοικονομικά ζητήματα. Ε, και είπε ότι για την ασφάλεια ε, θα πρέπει να δούμε και τι συνέπειες έχει για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και φυσικά αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η Γαλλία χρησιμοποιεί κάθε δυνατό επιχείρημα ε, προκειμένου να αποφύγει να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και να αποφύγει οποιαδήποτε συζήτηση και να δώσει περισσότερα ευρώ για τον προπολογισμό και βρισκόμαστε όμως σε αυτή τη ε, ε, θέση διότι τα θέματα ε, ασφάλειας και άμυνας να αποφασίζονται από τους Υπουργούς Οικονομικών νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει παρατραβήξει. Ορισμένες φορές ε, φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται καθόλου την ετοιμότητα των στρατιωτικών αστυνομικών δυνάμεών μας και των ε, υπηρεσιών πληροφοριών μας. Ένα σημείο με το οποίο θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Συνοχής που ανακύπτει συνεχώς σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις που κάνουμε τη σήμερα ημέρα είτε ε, αναφερόμαστε στην αναδιάρθρωση της νομισματικής ένωσης είτε ε, αναφερόμαστε σε προκλήσεις ε, που αφορούν την ε, μετανάστευση και τις απειλές της Ρωσίας ή πώς μπορούμε να διατηρήσουμε ασφαλή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αφορά το κατά πόσον μπορούμε να μείνουμε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι όταν δυσκολεύουν τα πράγματα και το να μείνουμε ενωμένοι ε, κυρίως ε, αφορά την τήρηση των συμφωνιών που έχουν ήδη συναυτεί. Επομένως, ε, το άρθρο 42, παράγραφος 7 και η όλη συζήτηση για το άρθρο αυτό είναι απλό έγινε εφαρμογή του. Όλα τα κρατημέλη συμφώνησαν ομόφωνα να αναγνωρίσουν το γεγονός αυτό και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένα να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην υπάρξει και νέα επίθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε καθηγητά. Θα ξεκινήσω τώρα με την ε, διαδικασία των ερωτήσεων. Θα ήθελα σας παρακαλώ όμως αγαπητοί συνάδελφοι να σηκώσετε χέρια όποιος θέλει να μιλήσει για να ελέγξουμε λίγο τον κατάλογο γιατί δεν είμαστε βέβαιοι. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση που έθεσα και σήμερα το πρωί. Κατά την εφαρμογή αυτού του άρθρου 42.7 ποιος ε, είναι ο αρμόδιος για να ελέγξει ότι όντω έχει υλοποιηθεί. Τα ίδια τα κράτη-μέλη που το επικαλούνται ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ότι εκπρόσωπο είναι αρμόδιοι ε, ε, δεδομένου ότι υπήρξε και ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει τι πρέπει να κάνει. Ε, τι πρέπει να γίνει, συγγνώμη. Ε, ε, το γεγονός ότι όλα τα κράτη-μέλη δέχθηκαν σημαίνει ότι αμέσως πρέπει να κινητοποιηθούν και να πούνε «Να, αυτά έχουμε». η γερμανική κυβέρνηση χρειάζεται έγκριση από το Bundestag, από τη Γερμανική Βουλή. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για να αιτιολογήσει τη δράση μεταξύ άλλων και για το 42-7. Σας διαβάζω αυτή τη ε, φράση στα γερμανικά. Η ε, καταπολέμηση του ISIS ως ε, δίκαιο ε, της ε, ε από το άρθρο 51 του ΟΗΕ του Συμβούλιο Ασφαλείου του ΟΗΕ περιλαμβάνει ότι όσον η συλλογική άμυνα για το καλό της Γαλλίας επιτυγχάνεται, τότε απαιτείται η συνεισφορά της Γερμανίας ε, του, μέσω του άρθρου 42.7 μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν είναι η νομική βάση με την οποία επέλεξε η γερμανική κυβέρνηση εσείς αναφερθήκατε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άρθρο το χρησιμοποίησε η, ε, η Γαλλία ούτως ώστε να αποφύγει ε, κάτι άλλο. Εμείς ως ε, αποφασίσαμε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσαμε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να αποφύγουμε το σύμφωνο σταθερότητας. Έχουμε ένα έγγραφο από τον συνάδελφο Κόντροβιτς και αυτή είναι η θέση μας Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι η δική σας αξιολόγηση ε, και αν το άρθρο 222 θα ήταν ίσως ε, μια καλύτερη λύση, ε, ένα καλύτερο άρθρο, διότι συγκεκριμένα αναφέρεται σε τρομοκρατικές επιθέσεις και αυτό ίσως θα έφερνε στο παιχνίδι καλύτερα ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Κάλερ. Ο κύριος Καν. Πολύ απλά κύριε Πρόεδρε, απλώς και κύριε καθηγητά, συγγνώμη, επειδή είστε εδώ και θα ήθελα να ξέρω το εξή. Αυτοί οι ε, ε οποίοι συνέγραψαν τη συνθήκη, τι ακριβώς είχαν κατά νου όταν έγραψαν αυτό το άρθρο, κύριο Μποστινάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσίασή σας, διότι αποδεικνύει ότι το περιεχόμενο του άρθρου, όπως έχει σχεδιαστεί από τη συνθήκη, με μία έκκληση για την εφαρμογή του μας έχει φέρει σε μία πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν ξέρουμε ποιος πρέπει να κάνει τι και πώς να συντονιστούμε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω δύο πράγματα. Ε, αναφερθήκατε σε κάποια από τα σημεία, αλλά νομίζω ότι η Σέγγεν χρειάζεται αποτελεσματικό έλεγχο συνόρων, όχι ένα, ε, έλεγχο στον οποίο τουλάχιστον ένα κράτος μέλος ε, θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι υπεράνω της ασφάλειας σε τέτοιες δραματικές περιπτώσεις Δεύτερον, μια βάση δεδομένων για να συλλέγουμε ή δυνατόν πληροφορίες ε, για τους τρομοκρατικούς κινδύνους και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη βάση αυτή όλα τα κράτη-μέλη. Κατόπιν, να υπάρχει πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών και όχι ε, πέντε με έξι χώρες ε, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και κάποιες άλλες να μην ανταλλάσσουν καν ή να κάνουν ε, ανταλλαγή πληροφοριών στη διακριτική τους ευχέρεια και να αποφασίζουν τι θα δώσουν σε ποιον και να έχουμε τρομοκράτες που θα πηγαίνουν έρχονται από το Παρίσι στο Βέλγιο και μετά στη Συρία και ποιος ξέρει που αλλού. Να υπάρχει λοιπόν πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών και όχι καταβούληση να υπάρχει μέσω ενός συστήματος το οποίο θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και συνεπές και επίσης να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών με εταίρους μας. ΝΑΤΟ, Ηνωμένε Πολιτείε, Ισραήλ, Αραβικό Σύνδεσμο, ε, κράτη του Αραβικού Συνδέσμου και το καθεξής. Αυτά πρέπει να γίνουν ώστε να προσδώσουμε μια κάποια ουσία στο άρθρο 42. Και τέλος, θεωρείτε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τα στοιχεία αποθεματικού τους ε, για την ε, ε, άμυνα, την ασφάλεια και να υπάρχει συμβατότητα και με το ΝΑΤΟ και να μην αποφεύγει και να ξεφεύγει από το ΝΑΤΟ γιατί αλλιώς θα πρέπει να μας δίνουν πληροφορίες οι ΗΠΑ γιατί εμείς από μόνοι μας δεν θα είμαστε σε θέση να συλλέξουμε πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στάνοκ. Θα ξεκινήσω με το θέμα που έθεσε ο κύριος Καν. Εγώ έχω αρκετή εμπειρία και είμαι ε, αρκετά ηλικιωμένος για να θυμάμαι από που ξεκίνησε το 1947. Ήταν δηλαδή πρωτοβουλία της Ελλάδας, επίμαχη θα έλεγα, και ουσιαστικά ενσωματώθηκε για να προστατεύσει την Ελλάδα αν υπήρχε πιθανή εισβολή στο Αιγαίο. Και βέβαια και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και ακριβώς γι' αυτό έχουμε την τελευταία παράγραφο που ουσιαστικά ε, δίνει υπεροχή στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Και αν το διαβάσετε και είστε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, είναι για μη στρατιωτική βοήθεια παρά για στρατιωτική. Είναι κάπως αδέξια βέβαια η διατύπωση στα αγγλικά και αμφίσιμη. Όμως η ερώτησή μου είναι διαφορετική ο όρος πόλεμος, γκέρ, όπως ε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εσείς φαίνεται να εθετείτε την έννοια αυτή ότι τα 28 κράτη-μέλη είναι σε πόλεμο με το Ισλαμικό κράτος, το ISIS. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε βεβαίως από νομική σκοπιά, γνωρίζοντας όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, Συζητήσαμε και τη Σύνοδο της Γενέβης, τη Σύμβαση της Γενέβης νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι τρομοκράτες του ISIS που κάνουν επιθέσεις, ε, αν συλληφθούν, θα είναι ε, κρατούμενοι πολέμου και θα πρέπει ουσιαστικά να τεθούν υποκράτηση σε τέτοιες συνθήκες. Δηλαδή τι είναι, γίνεται τελικά. Ε, μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, ο κύριος Μικέρ. Εγώ πρέπει ε, να πω ότι ε, μόλις τώρα ε, το Σαββατοκύριακο μίλησα το, με τον ιδρυτή του Ελεύθερου Συριακού Στρατού αλλά και με μια αραβική εκπομπή και αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι οι αεροπορικές επιθέσεις από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης ε, έχουν ε, κάνει ένα μεγάλο καλό ε, στους Άραβες και πάλι σε επιθέσεις που σκοτώνονται άμαχος πληθυσμός θα πρέπει λοιπόν ε, μέσω αεροπορικών επιθέσεων να ενισχύσουμε το μίσος του αραβικού πληθυσμού. Νομίζω ότι είναι αντιπαραγωγικό. Αλλά και αυτές οι αεροπορικές επιθέσεις ενισχύουν αντί να αποδυναμώνουν τον ISIS διότι γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η οργή του πληθυσμού και επιπρόσθετο, επιπρόσθετα υπόθηκε ότι θα πρέπει ε, τουλάχιστον να ανεχθούμε τον Ασάντ ε, και αυτό βέβαια θα αυξήσει ακόμα περισσότερο ε, την οργή του πληθυσμού με αποτέλεσμα έμεσα να ενισχυθεί επίσης ο ISIS. Θα πρέπει επίσης να είμαστε ε, πάρα πολύ ε, προσεκτικοί να συμπεριλάβουμε και το Ιράν σε αυτές τις στρατιωτικές σκέψεις διότι και εδώ, εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν, ε, υπήρχε αυτή η διαφωνία μεταξύ των Περσών και του αραβικού κόσμου. Έτσι λοιπόν τώρα με τις αεροπορικές επιθέσεις το να προσπαθούμε να θέσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση στην πραγματικότητα, δυσχεραίνουμε αντί να βελτιώνουμε την ε, κατάσταση, ενισχύουμε αντί να αποδυναμώνουμε τον ISIS. Ο επόμενος Τώρα το θέμα είναι πώς ε, θα χρησιμοποιηθεί ακριβώς αυτό το άρθρο. Η ερώτησή μου είναι ο εξή. Είπατε στην αρχή και σωστά ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ του 42.7 και του άρθρου 5 ότι το ένα ουσιαστικά έχει τις ικανότητες ενώ το άλλο όχι. Εγώ όμως θυμάμαι ότι ε, είχαμε το χάρη την διατύπωση τη Δικοευρωπαϊκής Συνθήκη για τη Δικοευρωπαϊκή Ένωση και εκεί το σχετικό άρθρο ήταν πιο ισχυρό από ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Υπήρχαν κάποιες ε, ερωτήσεις ε, αλλά και αναφέρθηκαν και σοβαρές αμφιβολίες. Εγώ θέλω να σας αναφέρω τώρα ποιες είναι οι αμφιβολίες μου. Ε, δεν ήταν για να αποκλειστεί η Ρωσία ή ήταν για να αποκλειστούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεύτερον, είναι αλήθεια αυτό που είπαν κάποιοι σχολιαστές ότι ο στόχος ήταν να ανακληθεί το σύμφωνο σταθερότητας γιατί εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει στη Γαλλία την Ιταλία, το Βέλγιο και η Αυστρία, ναι, για λόγους καταπολέμησης της τρομοκρατίας μπορείτε να έχετε μια άφεση. Έτσι λοιπόν ήδη λειτουργεί. Και η αμφιβολία μου είναι δεν ε, ζημιώνει το 42-7 γιατί κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί ίσως σε ένα απότερο μέλλον οι ικανότητες μπορεί να υπάρχουν και τότε θα έχουμε το άρθρο 5. Αλλά αν τώρα το μειώσουμε αυτό το άρθρο και το χρησιμοποιήσουμε έτσι ελαφρά την καρδία και ε, ουσιαστικά μετά την ε, Μαδρίτη ε, δεν μας είπατε γιατί δεν είχαμε το άρθρο 222 δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε το 322 ή το άρθρο 5 αν έχουμε μια επίθεση παρόμοια με τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου αλλά τώρα αν το χρησιμοποιούμε για πράγματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας ή όπως είπε ο κύριος Τάνοκ ότι είναι για μη στρατιωτικούς ε, σκοπούς Αν είναι δηλαδή κάτι τόσο αόριστο και δεν μιλάμε εδώ για, αμοιβαία, για ένα άρθρο αμοιβαία άμυνας για ρήτρα αμοιβαία έτσι όπως αποκαλείται ανέκαθεν, γιατί πρώτη φορά το επικαλούνται στην ιστορία, τι προσπαθώ να πω, ότι τελικά καταστρέφουμε το άθρος 42-7 εφόσον δεν το επικαλούμαστε στα πλαίσια της ορθής κατάστασης. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι που δεν ήταν παρόντες στην πρωινή συνεδρία τη Επιτροπής μας. Όπως θυμάμαι, το σημείο 6 είχε να κάνει με την ανταλλαγή απόψεων με τον του Γενικό Γραμματέα της Υπηρεσίας Εξωτερικές Δράσεις, τον κύριο Πέδρο Σεράνο. Και ένα από τα θέματα αφορούσε ακριβώς την ενεργοποίηση, την επίκληση αν θέλετε, του άρθρου 42.7. Ο κ. Σερένο μας ε, ενημέρωσε για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και σχετικά με την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παραγράφος 7 και μας είπε ότι η επίκληση του άρθρου αυτού είχε ως στόχο να ζητήσει την πιθανή βοήθεια με όλα τα μέσα σε διμερές επίπεδο από κάθε κράτος μέλος. Αυτά είναι τα γεγονότα. Αυτό μας είπε επίσημα ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Συγγνώμη, είμαι ήδη κουρασμένη. Παρακαλώ. Καθηγητά Μεπλερ, έκανα λάθος το όνομά σας. Σας ε, ευχαριστώ για το σύνολο των ερωτήσεων. Θα αναφερθώ πιο διεξοδικά σε ορισμένα θέματα. Κύριε Γκάλερ. Είπατε ποιος αξιολογεί τη συμμόρφωση. Αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με την ε, κάπως αβολή κατάσταση που έχει προκύψει σε ό,τι αφορά την απουσία μιας ε, επίσημης απόφασης του Συμβουλίου που μπορεί να έχει δώσει μια απάντηση σχετική. Δεν υπάρχει καμία όμως. Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το ποιος ε, θα αποφασίσει για το ποια είναι η επαρκής υποστήριξη. Και φαντάζομαι ότι η απουσία επίσημη απόφαση μα δείχνει ότι μπορεί να περιμένουμε ενδιαφέρουσε πολιτικέ συζητήσει στο μέλλον. Τώρα, αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θεωρηθεί ε, ως ένας τρόπος διεξόδου από το Σύμφωνο σταθερότητα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί πρέπει να πούμε το εξή. Μπορεί κάποιο να αυξήσει τις δαπάνες για την ασφάλεια χωρίς ε, να το κάνει αυτό ως τμήμα ενός προϋπολογισμού σε έλλειμμα. Απλώς ε, χρειάζεται να εξισορροπήσει σε αλλού τον προϋπολογισμό. Αλλά έτσι όπως ε, εκτελήσεται τώρα η διαδικασία μέσω διμερών επαφών και απουσία απόφασης του Συμβουλίου, απουσία θεσμικής συζήτησης για το τι σημαίνει το 42 παράγραφος 7, υπάρχει μια μπερδεμένη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές διαφωνίες εν τέλει. Επίσης, θέσατε το ερώτημα αν ε, το άρθρο 322 θα ήταν πιο κατάλληλο. Ναι και όχι, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εξαρτάται από το ποια πολιτική απάντηση θέλει να δώσει κανείς, τι απάντηση πολιτικής, το να επιλέξει το 427 δηλώνει ότι προτιμά μία απάντηση στρατιωτικού χαρακτήρα. Πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ που μας εξήγησε την ιστορική προέλευση του άρθρου αυτού της συνθήκης. Φυσικά κάποιος μπορεί να προσθέσει ότι υπάρχει προστιθέμενο ενδιαφέρον από κάποια κράτη-μέλη που μπορεί να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτό το άρθρο. Από τη δική του σκοπιά. Τώρα, σε σχέση με την ερώτησή σας. Εγώ δεν είχα σκοπό να στείλω το μήνυμα ότι είμαι υπέρ της ε, διατύπωσης αυτής ε, που χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με τον πόλεμο. Δηλαδή παρατηρώ ότι χρησιμοποιήθηκε. Ειλικρινά νομίζω ότι το μήνυμα θα ήταν πιο ισχυρό αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν ενώπιον του δικαστηρίου αντί απλώς ε, να σκοτωθούν σε μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση ή να, αυτό να την ακτούν. Τώρα να έρθω στην ερώτηση του κ. Μπούχνερ. Για το αν οι επιδρομές είναι μια επικοδομητική απάντηση. Υπάρχουν τα ορισμένα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Εγώ δεν θα προέβαινα σε μια σύγκριση μεταξύ των ρωσικών χτυπημάτων και των δυτικών αεροπονικών επιδρομών, γιατί είμαστε πολύ καλύτεροι από τους Ρώσους και ίσως οι Ρώσοι ε, μπορεί τελικά με τα χτυπήματά τους ε, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα γιατί ουσιαστικά θέλουν να στείλουν ένα στρατηγικό μήνυμα για το τι μπορούν να κάνουν θέλουν να στείλουν ένα τέτοιο μήνυμα στους γειτονές τους όμως η ουσία του ζητήματος είναι ότι υπάρχει μια στρατιωτική ισορροπία της εξουσίας ε, μεταξύ ποικιλών μερών. Θέλουμε εμείς να πλήξουμε, να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία υπέρ κάποιων μερών ή όχι προκειμένου να καταλήξουμε σε μια βελτιωμένη διπλωματική θέση. Αν η απάντηση είναι ναι, οι αεροπορικές επιδρομές μπορούν να παράσχουν μία απάντηση. Και κυρίως ό,τι αφορά την κατάσταση πέρσι, μια απαραίτητη απάντηση. Γιατί διαφορετικά μπορεί να είχαμε πετύχει Έτσι λοιπόν η αρνητική στόχη, δηλαδή μπορεί να είχε πέσει η Βαγδάτη είχαμε τον ενεργητικό στόχο να αποτρέψουμε να πέσει η Βαγδάτη στα χέρια του Ισλαμικού κράτους. Γιατί το θέμα που προσανατολίζει περισσότερο για το Ισλαμικό κράτος δεν είναι το γεγονός ότι κατόρθωσαν τελικά να ανατινάξουν κάτι. Αυτό είναι εύκολο εν τέλει. Αλλά το γεγονός ότι ουσιαστικά ασκεί το Ισλαμικό κράτος μια τέτοια γοητεία σε πολλούς νέους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει εδώ. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω των αεροπορικών επιδρομών. Και φυσικά όταν κάποιο προβαίνει σε αεροπορικέ επιδρομέ, θα πρέπει φυσικά να προσέχει και τι ακριβώ βαρδίζει. Κύριε Μποστινάρου. αναφέρεται ε, κάποια κέρια ζητήματα για το τι απαιτείται αυτή τη στιγμή με το χώρο Σέγγιν, αλλά θέλω να προσθέσω κάτι στη σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί από όσο γνωρίζω, ε, ουσιαστικά ανταλλάσσουν οι μυστικές, πληροφορίες, οι μυστικές υπηρεσίες πληροφορίες, δεν τις ε, μοιράζονται και ουσιαστικά ε, υπάρχει διευκόλυνση αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών, μάλλον της ανταλλαγή πληροφοριών, ε, με διάφορους τρόπους. Εσείς αναφέρετε τη βάση δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ισχυρό λόγο για το τι συμβαίνει με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Και αν πρέπει να βρεθούν κονδύλια, αν βρίσκονταν χρήματα, αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τις ε, μυστικές υπηρεσίες. Για τις υπηρεσίες πληροφοριών να εργαστούν προς κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις. Γιατί, ξέρετε, χρειάζονται μετρητά πολλές από αυτές τις υπηρεσίες. Και αυτό φυσικά μπορεί να γίνει κάλλιστα. Κατά κάποιο τρόπο ε, σκέφτηκα και την ταινία Edgar που ε, ουσιαστικά εξηγούσε πώς συστάθηκε το FBI. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών μετά το 13 Νοέμβρη. Και σε ό,τι αφορά τη διάστησή μου, πιστεύω ότι θα χρειαζόταν να έχουμε ένα και μόνο οργανισμό να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι αυτό κάτι στον ορίζοντα για το εγγύς μέλλον, ίσως. Αν και μιλώντας κοινικά, θα το πολιτικά δυνατό μόνο αν είχαμε περαιτέρω φορολογήσει. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για ολοκληρωμένε λύσει, το σημαντικό κομμάτι είναι να είμαστε ειλικρινεί για το τι θέλουμε και για το τι απαιτείται. Γιατί εξακολουθούμε ναι, να προσπαθούμε να κατανοήσουμε κάποιε από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες από την δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης. Ίσως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα πριν να συνεχίσουμε. Και κινδυνεύουμε να συνεχίσουμε κάνοντας τέτοια λάθη. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Κύριε Σαλουσκόφη, όσον αφορά το αν η συγκεκριμένη κατάσταση ε, αποτελεί ε, κινδυνό το άρθρο 42,7 να εφαρμοστεί και μελλοντικά. Ε, είναι πάρα πολύ νωρίς ε, να το κρίνουμε αυτό διότι μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε ποιο ακριβώς είναι το αποτέλεσμα. Ε, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνουν τα κράτη-μέλη ε, όσον αφορά αυτή τη λευκή επιταγή. Και σίγουρα βέβαια τα όσα θα προσφέρουν τώρα μπορεί να αλλάξουν στην πορεία. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα δούμε ε, μελλοντικά. Είναι ανοιχτό ακρό, ακόμα το θέμα. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι δεν αφορά τον αποκλεισμό μια οποιασδήποτε πλευρά, είτε πρόκειται για τη ΣΥΠΑ είτε για τη Ρωσία, αλλά πιο πολύ το ότι η Γαλλία νιώθει πιο άνετη ε, με ρυθμίσεις ε, που θα μπορεί, ε, στις οποίες θα μπορεί να έχει έναν ηγετικό ρόλο παρά το να Ε, όσον αφορά τουλάχιστον μια στρατιωτική επέμβαση παρά να παραδώσει ε, πλήρως ε, την ηγεσία σε κάποιον άλλο εταίρο διότι εν τέλει όταν κάνεις μια κοινή αεροπορική επίθεση εκστρατεία τότε αυτό πρέπει να γίνει κάπου οι αποστολές επικεντρώνονται κάπου και θα πρέπει όλο αυτό να γίνει με όλους τους παριστάμενους να έχει συζητηθεί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα πρώτο βήμα ούτω ώστε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή συνοπτική ανταπόκριση σε αυτό το θέμα ε, και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα ακριβώς να συζητήσουμε τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο πρόβλημα ασφαλείας προέκυψε και αυτό βέβαια συσχετίζεται και με το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας και αυτό δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού παρά μονάχα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά και τώρα θα ήθελα να ε, ζητήσω τη συμβουλή σας. Έχουμε ε, λίγο χρόνο ακόμα. Υποθετικά μπορεί να υπάρξει ένας δεύτερος ε, γύρος. Εγώ προσωπικά Αισθανόμαι ότι είχαμε αρκετό χρόνο ούτως ώστε να συζητήσουμε το άρθρο 42.7 αν επιθυμείτε μπορούμε να το ε, συνεχίσουμε όχι Οπότε θα ε, κλείσω αυτό το κομμάτι της ε, διάτεξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ματελέρ για τη συνεισφορά του ε, στη συγκεκριμένη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Now, any other business. Άλλα ζητήματα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω πού βρισκόμαστε όσον αφορά την απόφαση για, το, ε, για την Ολομέλεια σε δύο εβδομάδες Από την ε, πλευρά της ομάδας μου υποστηρίζω ότι θα ήθελα να έχω, θέλουμε να έχουμε μια συζήτηση και ε, προτείνω να εξετάσουμε ποια είναι η άποψη μεταξύ των ε, συναδέλφων για να προσθεθούν στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Είχαμε δύο ζητήματα της διάταξης τα οποία τα αφιερώσαμε σε αυτό το θέμα Κατά τη γνώμη μου αυτό το οποίο αναφέρθηκε από τον Πέτρο Σοράνο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη, ε, κατά τη δική μου γνώμη όμως ε, θα πρέπει να το προτιμήσουμε από το άρθρο 42.7 για παράδειγμα ή να προχωρήσουμε ε, περαιτέρω και να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτό και βέβαια ε, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για αυτό και σίγουρα μπορεί να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας Όμως νομίζω ότι υπό αυτές τις συνθήκες όπου δεν έχουμε ξεκάθαρες απόψεις ε, σχετικά με την ε, με τον σκοπό και την ε, νομική βάση για όλο αυτό και ε, καθώς επίσης και για τα περαιτέρω βήματα τα οποία θα ληφθούν από την πλευρά της Γαλλίας Νομίζω ότι επαφίεται στην Υποεπιτροπή να λάβει αυτόν τον ε, ρόλο, όμως αυτό το οποίο που μπορώ να προτείνω εγώ είναι ότι θα πρέπει ε, το πολιτικό έργο να το ξεκινήσει αυτό. Αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου γνώμη. Προσκαλώ βέβαια τους συναδέλφους να το συζητήσουμε κύριε Χάν ε, θα ήθελα να πω ότι θα το εξετάσουμε αυτό στην ομάδα μας Άλλα μέλη. Κύριε Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να πω ότι παραμένω ε, σκεπτικιστής όσον αφορά αυτήν την ιδέα. Η συζήτηση σήμερα ήταν πιο ακαδημαϊκής φύσεως και θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Διότι Εν τέλει, αυτό σημαίνει ότι ο διακυβερνητικός μηχανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εμείς έχουμε βέβαια λόγο ως κοινοβούλιο και έχουμε μια λειτουργία ε, ε, επίβλεψης ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή την ακαδημαϊκή συζήτηση. για να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει ε, κάποιο πέρδεμα. Εμείς θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Άλλες πολιτικές ομάδες Πιστεύω ότι μία συζήτηση είναι κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Το τι αποτέλεσμα θα υπάρξει είναι κάτι ε, θα πούμε αυτό το οποίο θα το δούμε αυτό που πρότεινε ο κ. Γκέλα ε, θα πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί. Αυτά τα οποία είπα σχετικά με την ε, πιθανή απόφαση δεν σημαίνει ότι ε, θα υπάρξει συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ε, συζητούμε σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ψήφισμα θα πρέπει να συζητηθεί στις επιτροπές. Ή όπως ε, ήθιστε, αν θα υπάρξει ένας, μια πολιτική συζήτηση μία από τις πολιτικές ομάδες ε, θα πάρει την ε, πρωτοβουλία και ίσως να οδηγήσει τελικά σε έναν ε, συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων που εν τέλει θα οδηγήσει σε ένα σχέδιο ψηφίσματος. Δεν βλέπω λοιπόν λόγο για, γιατί η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει ως εκεί. Όμως η χώρα που για πρώτη φορά ενεργοποίησε το άρθρο 42.7 ήταν αυτή ακριβώς η ιδέα της να συνεχίσει τη διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο και κατά τη γνώμη μου λοιπόν ε, δεν χρειάζεται κάποια άλλη διαδικασία αυτή η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε αυτό το κοινοβούλιο ως πρόεδρος της υποεπιτροπής λοιπόν θα πρότεινα εάν οι ε, ομάδες συμφωνούς αυτό δεν θα είναι πρωτοβουλία της υποεπιτροπής. Ήταν ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο ε, επικεφαλής της ομάδας εξωτερικών υποθέσεων ε, είπε στην δική μας υποεπιτροπή να ασχοληθούμε με αυτό και το ότι θα πρέπει ίσως να υπάρχει μια τέτοια ε, πρωτοβουλία από εμάς που θα οδηγήσει σε ψήφισμα και δεν λέω ότι, θα γράψω τώρα μια θέση, ένα, ε, μια εργασία σχετικά με τον σκοπό της 42α, 42 α 42 εφτάσει. Και πιστεύω λοιπόν ότι όσο ασχολείται με αυτό το θέμα ένα θέμα το οποίο ε, έρχεται στο πλαίσιό μας ε, και θα πρέπει να αφήσουμε άλλες επιτροπές, υποεπιτροπές να κάνουν τη δική τους δουλειά και να την παρουσιάσουν στο Κοινοβούλιο και, και το θέμα είναι αυτό ότι οτιδήποτε ε, είναι δική μας εντολή θα πρέπει να οδηγηθεί στην Ολομέλεια και έχει υποστηριχθεί από την ομάδα των σοσιαλιστών ε, και από τους ε, πράσινους, οπότε έχουμε μια πλειοψηφία να το θέσουμε. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα σκοπό να παρέμβω διότι εγώ είμαι προσκεκλημένος σήμερα, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Ασφάλεια και Έμενα. είμαι μέλος ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά ε, μιλώ εξ ονόματος της ομάδας μου, της Ευρώπης των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, όπως είστε και εσεί μέλο τη ομάδας, κυρία Φωτίγκα, και νομίζω ότι θα πρέπει να παρέμβω για την θηγατρική επιτροπή, διότι η ε, επιτροπή σας είναι η επιτροπή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Η ομάδα μου λοιπόν θα ανησυχήσει ιδιαίτερα αν σκοπός αυτής της διαδικασίας ήταν να γίνει κάποια επιτροπή θεματοφύλακα των συνθήκων για να επιβλέψει την εφαρμογή του 42-7 ή οτιδήποτε θέλει να περάσει τη διαδικασία στην Επιτροπή ε, της Αμοιβαίας συλλογική άμυνας. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στην ε, στο ΝΑΤΟ και στο γεγονός ότι προτεύει το ΝΑΤΟ, όπως άλλωστε ε, προβλέπεται και στη διαδικασία αν πρόκειται για θέμα ασφάλειας και άμυνας και δεν θα ήθελα να υπάρχει κάποιο ψήφισμα το οποίο θα ε, σημαίνει ότι υφαρπάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής την αρμοδιότητα για την ε, ε σύγκληση και την εφαρμογή του άρθρου 47 42-7. Μιλώ εξ ονόματο της ομάδας μου σε επίπεδο επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και δεν είναι εδώ νηστή μα σήμερα. Κύριε Γκάλερ, ε, νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Προσπάθησα να το επιλύσω λίγο ε, με διπλωματικό τρόπο, λέγοντας ότι η κατάσταση αυτή, κατά την άποψή μου, ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ε, είμαστε αλληλέγγυοι προς τη Γαλλία. Το έχουμε κάνει επανειλημμένως, το κάναμε και στην προηγούμενη Ολομέλεια. Το θέμα αυτό δεν αφορά όμως ε, θέμα μόνο την αλληλεγγύη προς τη Γαλλία, διότι η Γαλλία θέλησε να προχωρήσει σε διμερές επίπεδα με τα κράτη-μέλη. Επομένως, κατά την άποψή μου, αυτό υπερβαίνει την ε, επιθυμία της χώρας ε, που επικαλείται τη χρήση του άρθρου 42.7. Εγώ δεν ήμουν παρούσα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ζητώ συγγνώμη την έχασα αυτή την ε, δήλωση που αναθέτει στη ΣΕΝΤΕ να προχωρήσει το ψήφισμα, αλλά νομίζω ούτως ή άλλως όλοι έχουμε μία ελεύθερη εντολή και δεν ε, ε, το συζητήσαμε στο διευρυμένο Προεδρείο, μπορούμε να το κάνουμε βέβαια. Το είχαμε προγραμματίσει για τη Σύνοδο της Ολομέλειας, συζητήθηκε στη διάρκεια της Ολομέλειας λοιπόν της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. και μάλιστα ε, είχαμε δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης τα οποία τα συζητήσαμε συνολικά πάνω από δύο ώρες συζητήσαμε και το περιεχόμενο και τις πιθανές συνέπειες ε, της εφαρμογής του άρθρου 42.7 και νομίζω ότι βάσει αυτής της συζήτησης δεν συντρέχουν και τόσοι νομικοί λόγοι για μία λύση που ε, θα υπερβαίνει τα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου και πολύ σωστά εξήγησε και ο κύριος Σεράνο, Σοράνο ότι αυτό είναι στα πλαίσια της αμοδιότητας των κυβερνήσεων ε, και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία που υπέδειξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καλό θα ήταν να συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο, να το συζητήσουν οι πολιτικές ομάδες, ε, να προσπαθήσουν να βρουν μια συνένεση και να συμφωνήσουν. Ο κύριος ε, Έλερ. Σχετικά με τα όσα είπε ο κύριος ε, Τένοκ, ε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, μπορεί να γίνει ένα τέτοιο αίτημα και αυτό το οποίο είπατε εσείς ε, είναι μια ακαδημαϊκή, ένας ακαδημαϊκός σχολιασμός των όσων συζητήθηκε. Όταν λοιπόν οι δύο μεγάλες παρατάξεις κάνουν μια αίτηση τότε πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό και στο πλαίσιο της ε, συζήτησης ε, μπορεί να υπάρχει η ίδια ή διαφορετική πολιτική άποψη ε, και η ίδια ακαδημαϊκή άποψη, όμως κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρξει μια πρόσφαση, πρόταση ψηφίσματος και όχι μια συζήτηση. Εντάξει λοιπόν, Σίγουρα υπάρχει διαδικασία. Αυτό το οποίο έλεγα εγώ όμως είναι ότι με βάση τις συζητήσεις μας δεν είναι τόσο σαφή τα πράγματα ώστε να αναλάβει ένα επίσημο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα ενία στο θέμα αυτό. διότι δεν υπάρχει ακόμα ε, παρακολούθηση του θέματος από... δεν έχει δοθεί συνέχεια συγγνώμη, από τα κράτη-μέλη, δεν έχει συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο και αυτό ε, είναι η άποψή μου. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι οι δύο πολιτικές ομάδες ε, θέλουν ε, να προωθήσουν το ζήτημα αυτό και να το κάνει η Επιτροπή μας, αλλά ε, προς το παρόν θα ήθελα να σταματήσει εδώ η συζήτηση Θα επικοινωνήσω και θα σας ανακοινώσω την απόφασή μου. Ε, συνεδριάζουμε την Πέμπτη ούτως ή άλλως. Μέχρι τότε μπορούμε να βρούμε μια λύση, λέει ο κύριος Γκέλλερ. Ναι, να πω απλώς ότι την Πέμπτη έχουμε μια κοινή έκτακτη συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο θα γίνει από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ και υπάρχει ένα δεύτερο σημείο που είναι ξεχωριστά μόνο για την Επιτροπή μας και είναι για την ακρόαση για, με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας. Πέρα στη συνεδρία, σε ευχαριστώ πολύ.